Καλημέρα συνάδελφοι, ξεκινάμε τη συνεδρίαση. Θα περάσω στην Ιταλική γλώσσα. Το πρώτο θέμα είναι οι αποφάσεις που ελήφθησαν χθε το απόγευμα από τους συντονιστές. Οι συντονιστές έλαβαν υπόψη την εφαρμογή των μεθόδων εργασίας της Επιτροπής Αναφορών χάρη στο συνθετικό κείμενο το οποίο προετοίμασε η Γραμματεία επί του εγγράφου αυτού και επί των αποτελεσμάτων του εγγράφου αυτού οι συντονιστές αποφάσισαν να υπάρξει ένας περιοδικός έλεγχος και να ενημερώνονται και να εμπλουτίζονται το κείμενο αυτό σύμφωνα με τους νέους κανόνες που υιοθετήσαμε τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2013 λάβαμε υπόψη μας ε, οι συντονιστές τα θέματα που αφορούν την μελλοντική ε, ε, θύρα στο διαδίκτυο και γι' αυτό θα προετοιμαστεί ένα κείμενο το οποίο θα επιτρέψει να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις όπως ακριβώς έχει προταθεί επανειλημμένα από την συνάδελφη Άουκεν σεβόμενοι τους κανόνες και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Οι συντονιστές ενέκριναν επίσης το αίτημα για μια ειδική έκθεση που ζήτησε η διαμεσολαβήτρια για το θέμα του ελέγχου των εξουσιών του Frontex και επί των κατεπηγουσών διαδικασιών απερίψαν οι συντονιστές τις ψηφοφορίες τις ομαδικές και ζήτησαν να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά τα διάφορα αιτήματα με μεμονωμένο δηλαδή τρόπο. Για τις δέκα αναφορές οι οποίες έχουν σχέση με το θέμα της ρύθμισης των μεταναστευτικών ρευμάτων στην Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα το θέμα της Λαμπεντούζα, οι συντονιστές ε, ψήφισαν ομόφωνα για τη χρήση της διαδικασίας του κατεπήγοντος. Για το θέμα το οποίο αφορά την, το αίτημα την αναφορά Γκαλαντίνο για την πιθανή παραβίαση των αρχών της αναδρομικότητας και της νομιμότητας σχετικά με την εφαρμογή του Ιταλικού νόμου 109 του 12 Απέριψαν την χρήση της κατεπίγουσας διαδικασίας γιατί δεν έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες αυτά τα νομικά κείμενα. Για την αναφορά του κυρίου Τσίτσεστερ για μια κατεπίγουσα διαδικασία σχετικά με το πρόβλημα ε, της συνοριακής σύνδεσης Ισπανίας και ε, Γιβραλτάρ απέρριψαν οι συντονιστές τη διαδικασία κατεπίγοντος, θεωρώντας απλά ότι δεν είναι κατεπήγον το θέμα. Απέριψαν επίσης και το αίτημα Μπέκερ ε, για την ασφάλεια στους πυρηνικούς ευρωπαϊκούς αντιδραστήρες ε, με πλειοψηφία και ομόφωνα δέχθηκαν το αίτημα Μπουλάντ ε, ε, σχετικά με την απέλαση του κυρίου Τζιλμπέρτη. Για την ημερήσια διάταξη οι συντονιστές θα ε, καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους με την διανομή των αποφάσεων γραπτά, κάτι το οποίο δεν έγινε ε, χτες και θα γίνει στην επόμενη συνάντηση στις αρχές Δεκεμβρίου. Σχετικά τώρα με τις συστάσεις που έκαναν ορισμένοι συνάδελφοι γύρω από τις αναφορές. Έγινε ομόφωνα δεχθεί η γνωμοδότηση για τις τροποποιήσεις ε, για όλα τα αιτήματα που είχαν κατατεθεί εκτός από το τελευταίο όπως ακριβώς ε, θα φανεί και στα πρακτικά ταυτόχρονα έγιναν κάποιες επιπλέον ανακοινώσεις ε, χαρακτήρα, που έχουν χαρακτήρα τεκμηρίου θα έλεγα και είναι διαθέσιμα στη γραμματεία και διαθέσιμα στη διάθεση όλων σας. Υπάρχει ένα επιπλέον θέμα το οποίο αφορά την έκθεση για την Γαλλικία το οποίο είναι το σημείο 16 για σήμερα. Χθε ψηφίσαμε την τροποποίηση της ημερησίας διατάξεως, ακυρώνοντας το θέμα αυτό. Οι συντονιστές αποφάσισαν όμως ότι η έκθεση θα επανεξεταστεί σε μία συνάντηση την οποία θα προετοιμάσει ε, το Προεδρείο της Επιτροπής έτσι ώστε να υπάρξει μία συμφωνία ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής ως προς το ε, περιγραφικό τμήμα θα έλεγα και επιβεβαίωσαν το χρονοδιάγραμμα για την ψηφοφορία της συγκεκριμένης εκθέσεως, 17 κατάθεση τροπολογιών, 5 συζητήσεις, 16 ψηφοφορία και από εκεί και πέρα ε, δεν αποφασίστηκε κάτι άλλο από πλευρά των συντονιστών. Ε, αυτές ήταν οι αποφάσεις τους, γίνονται ελπίζω δεκτές και περνώ στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Δεν υπάρχουν ε, λοιπόν διαφωνίες και περνάμε τώρα στο σημείο 15. Punto 15 che è la relazione 2013 sulla cittadinanza. Η έκθεση 2013 για την ηθαγένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγητής είναι ο συνάδελφος κύριος Σαλαβράκος, τον οποίο θα δώσω αμέσω το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, και συνάδελφοι, η έκθεση βασίζεται στην αρχή ότι κάθε άτομο με ηθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και Ευρωπαίος πολίτης Η έκθεση βασίζεται στην αρχή ότι κάθε άτομο με ηθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και Ευρωπαίος πολίτης. Επομένως η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρώνει χωρίς να αντικαθιστά την εθνική ηθαγένεια. Γι' αυτό και το δικαιώματα των πολιτών αποτελούν κύριο γνώμονα της έκθεσης και το δικαίωμα προσφυγής των διαμεσολαβητή, το δικαίωμα υποβολής νομοθετικών προτάσεων με πρωτοβουλία πολιτών, καθώς και το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεσαι στις δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές αποτελούν σημαντικά και αναπόσπαστα δικαιώματα των πολιτών. Ο συζητητής της έκθεσης σχετικά με την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013 και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών θεωρώ ότι είναι σημαντικό να σας αναφέρω κάποια σημεία της εκθέσεως που αναδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους. Είναι σημαντικό τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών να κατοχυρώνονται και να περιγράφονται σαφώς από τις νομικές προβλέψεις της Ένωσης και να εφαρμόζονται έτσι ώστε οι πολίτες να νιώθουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζω λοιπόν ότι το δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, δημιουργώντας ένα διάβλο επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, και μετατρέποντας την Ένωση σε μια σημαντική έννοια για τους πολίτες της. Η δημόσια εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Οι ευρωπαϊκές εκλογές πρέπει να στοχεύσουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών στο πολιτικό σύστημα και στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας. Οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις συνθήκες ώστε να έχουν καλύτερη κατανόηση για τα πρακτικά ωφέλη της ευρωπαϊκής σταγένειας. Η Επιτροπή Αναφορών προσπαθεί να διορθώσει αυτά τα προβλήματα θέτοντας τους πολίτες στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους το νέο One Portal της Επιτροπής Αναφορών το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις αρχές του 2014 θα μετατρέψει τη διαδικασία αναφορών σε ένα ελκυστικό και εύχριστο μέσο. Η απόκτηση και η απώλεια της ταγένειας των κρατών μελών ρυθμίζονται αποκλειστικά βάσει του εθνικού δικαίου των επιμέρους κρατών μελών και βάσει της αρχής της επικουρικότητας. Είναι σημαντικό να μην παραβλέψουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικέ ανάγκες που θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. Ε, είναι βασικά σημεία της εκθέσεως και δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Πιστεύω ότι ήδη ε, έχετε κάνει μια πρώτη ανάγνωση. Ε, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Μοντέλο βρίσκονται σε μια δύσκολη καμπή τόσο της αξιοπιστίας τους όσο και των οικονομικών προοπτικών της Ένωσης συνεπία της οικονομικής κρίσης γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια στους Ευρωπαίους πολίτες. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είναι έτσι. Πρέπει να αποδείξουμε ότι ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο όλης της φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευελπιστώ ότι θα κατορθώσουμε να εφαρμόσουμε την αρχή αυτή. Κλείνοντας, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων πάνω σε αυτά τα οποία ανέφερα, καθώς και σε όλα τα θέματα που πιθανόν θεωρούν σημαντικά για να αναπτυχθούν μέσα από την έκθεση και θα περιμένω με χαρά τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Σαλαβράκο. Η κυρία Σντάνοκα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων προς τον κύριο Σαλαβράκο. γιατί παρουσίασε πάρα πολλές χρήσιμες συστάσεις στην έκθεσή του και υποστηρίζω πλήρως αυτά τα οποία λέγονται στο κείμενο. Να μου επιτρέψετε όμως να προσθέσω κάποια επιπλέον σημεία αν θέλετε ή να ζητήσω εν πάση περιπτώσει να υπογραμμιστούν κάποια σημεία που ήδη περιλαμβάνονται στην έκθεση. Όταν μιλάμε για αυτή την ευρωπαϊκή ιδιότητα που είναι και η χρονιά της φέτος. Και μιας και προετοιμάζεται μια νέα κατάσταση γύρω από αυτό, με φοβίζει θα έλεγα μια στενή ερμηνεία του φαινομένου αυτού που αφορά αποκλειστικά την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών και που βάζει στην άκρη αν θέλετε, ένα σημαντικό παράγοντα της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος δεν περνάει από τη μία χώρα στην άλλη μόνο και μόνο για να ταξιδέψει για οικογενειακούς λόγους, αλλά αναφέρομαι στους εργαζομένους ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελεύθερη δυνατότητα εγκατάστασής τους σε άλλες χώρες με πλήρη δικαιώματα και συμπεριλαμβάνονται εδώ τα κοινωνικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσώπων, το δικαίωμα στην αντικατάσταση των κοινωνικών παροχών που είχαν κάποτε στην καινούρια χώρα, συνταξιοδοτικά δικαιώματα και αναγνώρισή τους κτλ. Εδώ ε, τα θέματα χαίνουν, τα είναι πάρα πολύ σοβαρά, ε, παίρνουμε και εμείς πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα μη σεβασμού των δικαιωμάτων μέσω των αναφορών και πρέπει να αντιμετωπιστούν με το σωστό τρόπο και να συμπεριληφθούν φυσικά και στην έκθεση. Έχουμε πάρει πάρα πολλές αναφορές για την αναγνώριση των πτυχίων, σαν παράδειγμα των επαγγελματικών προσόντων κτλ. Κάτι άλλο το οποίο περιλαμβάνεται ε, στην έκθεση αλλά θα ήθελα να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο είναι το θέμα της διπλής υπηκότητας και την απώλεια της υπηκότητας σε μία χώρα λόγω της απόκτησης μιας υπηκότητας σε, άλλο χώρο, σε άλλη χώρα συγγνώμη, Έχετε ακούσει τις περιπτώσεις της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας λοιπά μέσω ε, αναφορών που έχουν κατατεθεί. Το πρόβλημα ε, το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι ότι η υπηκότητα του Ευρωπαίου πολίτη δεν προσφέρει στην παρούσα φάση προστιθέμενη αξία. Είναι ένα παραγόμενο δίκαιο της ε, ιδιότητας του, του πολίτη της κάθε χώρας. Και υπάρχουν δύο απόψεις επ' αυτού. Η μία η οποία το αντιμετωπίζει αυτήρα πολιτικά και λέει ότι η ευρωπαϊκή υπηκότητα θα πρέπει να παρουσιάζει κάποια δυνατότητα προστιθέμενης αξίας και να την δημιουργεί και μια άλλη άποψη η οποία λέει ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να υπάρχει και πρέπει να είναι ουδέτερη. Η προστιθέμενη αυτή αξία λοιπόν θα πρέπει να περιλαμβάνει σαν παράδειγμα την δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι πολίτες της χώρας στην οποία πηγαίνουν. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια οδηγία η οποία καλύπτει με ξεχωριστό τρόπο και δίδει κάποια δικαιώματα στους πολίτες αυτούς, αλλά δεν τους αποδίδει πλήρη δικαιώματα όπως έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες γενικά στην κάθε χώρα. Υπάρχει μάλιστα μία ομάδα και σε αυτούς τους πολίτες από τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν έχουν καμία ιδιότητα πολίτη από καμία χώρα, καμία υπηκότητα. Είναι οι λεγόμενοι μη πολίτες της Λετωνίας και οι μη πολίτες της Εσθονίας. Έχουμε κάποιες αναφορές από την Εσθονία για τη δυνατότητά τους να παίρνουν μέρος στις ευρωπαϊκές εκλογές. Έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν οι πολίτες αυτοί στις τοπικές εκλογές και θέλουν να πάρουν μέρος και στις ευρωπαϊκές εκλογές. Έχουμε πάρει μια αναφορά με 16.000 υπογραφές και από τη Λετωνία, όπου οι λεγόμενοι μη πολίτες δεν έχουν κανένα εκλογικό δικαιώμα σε καμία εκλογή είτε ε, τοπική, είτε περιφερειακή, είτε ευρωπαϊκή. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν προτάσεις που να ενισχύουν τα δικαιώματα των πολιτών και τα δικαιώματα των πολιτών να επεκτείνονται σε όλους τους πολίτες μιας χώρας. Θα πρέπει νομίζω αυτό να γίνει αντικείμενο αναφοράς στην συγκεκριμένη έκθεση. Να προσθέσω κάτι επιπλέον το θέμα της διπλής υπηκότητας που δεν γίνεται αποδεκτή από τις νομοθετικές ρυθμίσεις κάποιων χωρών. Οι περιπτώσεις ε, των Ούγκρων της Σλοβακίας, σαν παράδειγμα, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αν η ευρωπαϊκή ιδιότητα παρουσίαζε ακριβώς αυτήν την επιπλέον αξία αν είχαν την ευρωπαϊκή υπηκότητα την οποία δεν μπορούν να απολέσουν τότε θα είχε επιληθεί το θέμα. Γνωρίζω βέβαια ότι υπάρχουν ε, διστάμενες απόψεις, υπάρχουν ε, διαφορετικές πολιτικές προτάσεις γύρω από το θέμα αυτό. Παρόλα αυτά νομίζω ότι θα παρουσίαζε ενδιαφέρον για μας, για Επιτροπή Αναφορών, να αντιμετωπίσουμε το θέμα ε, μιας και έχουν κατατεθεί αρκετές αναφορές σχετικά με το θέμα της διπλής υπηκότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καθώς επίσης ευχαριστώ και τον εισηγητή κύριο Σαλαβράκο. Βλέπω στην έκθεση αυτή ένα πραγματικά ισορροπημένο έργο και είμαι πεπισμένος ότι μπορώ να παρακινήσω και τους συναδέλφους μου του Λαϊκού Κόμματος να την υποστηρίξουν. Πολύ θετικά την κρίνω. Έχω ορισμένα σχόλια προς μια, ποια κατεύθυνση μπορώ να φανταστώ ότι ίσως υπάρχει χώρος βελτιώσεως. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην τελευταία έκθεση προτείνονταν 25 μέτρα από την Κομισιόν. Είχαν μάλιστα ανακοινωθεί και τα περισσότερα εφαρμόστηκαν. Αυτό είναι θετικό. Επίσης, ο ρόλος της ενιαίας αγοράς με την ενίσχυση των καταναλωτών επίσης εντάσσεται εδώ σε μια προσπάθεια δηλαδή τόνωσης της σημασίας της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Υπάρχουν λοιπόν πολλές θετικές πτυχές όπως και η σχετική δικτυακή, πύλη. Είμαι εισηγητής του Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή πολιτισμού. Εκεί θα αναπτύξω στη δική μου γνωμοδότηση κάποιες απόψεις με στόχο ώστε η συνείδηση του Ευρωπαίου πολίτη καθώς επίσης και η γνώση για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια να περιληφθεί στη μελλοντική εκπαιδευτική πολιτική. Θέλω να τονιστεί η σημασία της ευρωπαϊκής εκπαιδεύσεως. Στι δικέ μου τροπολογίε που θα υποβάλω στην Επιτροπή Αναφορών επιθυμώ να τονίσω ιδίω την ανάγκη ενίσχυση των πολιτικών δικαιωμάτων καθώς επίσης και την στράτευση των πολιτών σε μη κρατικέ οργανώσεις, σε εκκλησίες κλπ. Χρειαζόμαστε εντό εισαγωγικών ιεραποστόλους οι οποίοι θα φέρουν πολύ πιο κοντά στο πνεύμα και στη διανόηση των Ευρωπαίων την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια βρίσκω και πάλι εξαιρετικά θετική την έκθεση και θα την χειριστώ με τον τρόπο που σας είπα, τη δική μου πλευρά δηλαδή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση του συναδέλφου του κυρίου Σαλαβράκου είναι πάρα πολύ σημαντική διότι με αφορμή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη και το θέμα του πολίτη της Ευρώπης ποιος είναι ο πολίτης της Ευρώπης, αλλά και με αφορμή πάμπολες αναφορές που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θίγουν ή διεκδικούν τα δικαιώματα των πολιτών, η έκθεση πράγματι πρέπει να ακουμπάει στην πραγματική κατάσταση σήμερα. Με αυτή την έννοια ε, είναι σοβαρή η διεκδικουν τα δικαιωματα των πολιτων η εκθεση πραγματι πρεπει να ακουμπαει στην πραγματικη κατασταση σημερα με αυτη την εννοια ειναι σοβαρη η δουλεια που έκανε ο κύριος Σαλαβράκος. Οι δικές μου παρατηρήσεις αφορούν θέματα που έχουν σχέση με την ίδια την ταυτότητα και νομικά ας πούμε, την ηθαγένεια, αλλά κυρίως με τα δικαιώματα των πολιτών. Σημείο πρώτο δηλαδή που θέλω να πω. Καταγράφεται και σε το δικό μας το κείμενο, θα λέγεται και λέγεται με πολύ άνεση ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι στις ευρωεκλογές πιθανόν να έχουμε μεγάλα ποσοστά αποχής. Αλλά εδώ αυτή η διαπίστωση πρέπει να εξηγηθεί και κατά τη γνώμη μου και δεν είναι πια γνώμη μου φαίνεται από τις μετρήσεις τουλάχιστον στις χώρες του Νότου με τις ακολουθούμενες πολιτικές της λιτότητας τις σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές ο πολίτης γιατί ο πολίτης είναι και εργαζόμενος δεν είναι απλά δικαιώματα πολιτικά αισθάνεται μακριά από αυτή την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυσφορεί με αυτές τις πολιτικές. Πρώτον λοιπόν το να εξηγούμε ότι το να λέμε ότι θα υπάρχει χαμηλή συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες των ευρωεκλογών δεν απαντάμε στο πρόβλημα. Θα μου πείτε η έκθεσή μας έχει τέτοιο χαρακτήρα. Θα έλεγα ναι. Για την πληρότητα ναι. Θα πρέπει να εξηγήσει γιατί βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο. Το οποίο δυστυχώς αν συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές θα συνεχιστεί. Θα διευρυνθεί μαζί με άλλα παρεπόμενα φαινόμενα που και αυτά είναι θέματα τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Το δεύτερο, εδώ έχει δίκιο ο κύριος Αλαβράκος ε, ενώ το πρώτο θεωρώ ότι θα μπορούσε να το συμπληρώσει, δεν περιέχεται η πρώτη διαπίστωση. Στο δεύτερο σημείο που θέλω να σταθώ είναι ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει πιο δημοκρατική και πιο ανοιχτή στους πολίτες. Είναι σωστή αυτή η επιστήμανση και εννοώ τις διαδικασίες και όλα αυτά. Εμείς έχουμε μια αίσθηση όσο αφορά το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες την Επιτροπή μας ως ένα δείγμα. Νομίζω ότι εδώ πράγματι πρέπει να τονιστεί ακόμα περισσότερο το σημείο αυτό, ιδιαίτερα ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο, ο μόνος ερετός θεσμός στο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατήρηση τρίτη, υπάρχει με τα δικαιώματα των το θέμα των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών που μετακινούνται σε άλλη χώρα, από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θα πρέπει να δούμε πώς διατηρούν το δικαίωμα να ψηφίζουν και στη χώρα προέλευσης ή για τη χώρα προέλευσης, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες για της ψηφοφορία, από τη χώρα υποδοχής για τη χώρα προέλευσης. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να επισημανθεί και που σαφώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ δεν νομίζω ότι θα έχουμε ε, πρόβλημα. Απλώς επισημαίνω ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι οριακό καθώς τουλάχιστον από τη πατρίδα μου αλλά και από άλλες χώρες θα επαναλάβω του Νότου έχουμε νέους μετανάστες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξέβρεση εργασίας που πιθανόν αυτό θα να σημαίνει μακροχρόνια παραμονή τους εκεί για τους λόγους για τους οποίους αναζητούν ε, εργασία. Τέταρτο σημείο, εδώ συμφωνώ ότι πρέπει να απλοποιηθούν οι, συνθήκες για να ευκολύνονται, να οι μετακινήσεις μεταξύ των πολιτών της Ένωσης. Σας επισημαίνω αγαπητοί συνάδελφοι από την εμπειρία άλλων επιτροπών ότι στον ορίζοντα δεν είναι κάτι σαφές, απλώς το λέω ε, έρχονται περιορισμοί μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους επιλεκτικής στάσης που κρατάνε ορισμένες χώρες όσο αφορά τους εργαζόμενους. Να το επαναλάβω με πιο απλά λόγια, δεν είναι εύκολη ή δεν θα είναι εύκολη η μετακίνηση ενός εργαζομένου ας πούμε από την Ελλάδα, μηχανικού, γιατρού, τον οποίον ζητάει τώρα η Γερμανία και αύριο δεν θα το θέλει. Στον ορίζοντα έχω ακούσει και σχέδια να μην έχει τέτοιες τέτοια δυνατότητα ελεύθερη μετακίνηση Και το επισημαίνω διότι πρέπει να κατοχυρωθεί. Και πρέπει να κατοχυρωθεί και με συγχωρείτε που λέω παραπάνω, διότι είναι ένα από τα βασικά κριτήρια στο κατά πόσον φτιάξαμε έναν ενιαίο χώρο, που είναι η ελευθερία και η κινητικότητα των εργαζομένων. Η κινητικότητα τη εργασία. Επομένω είναι από τα βασικά δικαιώματα έτσι όπω θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τι τέσσερι ελευθερίε για όσου του αρέσουν να παραπέμπουμε στι ελευθερίε αυτέ. Επομένω υπάρχει ένα πρόβλημα αυτό και ένα δεύτερο όταν έρχονται άνθρωποι από άλλες χώρες εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα για την κατοχήρωση των δικαιωμάτων. Μιλώ για τους μετανάστες. Είμαστε αντίθετοι, όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Αριστερά με τη συνθήκη της Λισαβόνα. Είμαστε αντίθετοι διότι, κατά τη γνώμη μας, ουσιαστικά στα θέματα αυτά κάνει την Ευρώπη Ευρώπη φρούρη. Εδώ πρέπει στο επίπεδο των δικαιωμάτων, γιατί ανοίξαμε τέτοια θέματα και σωστά ανοίγει θέματα τέτοια η έκθεση, οι διαδικασίες απόκτησης της ηθαγένειας των μεταναστών αλλά και των παιδιών τους που γεννιούνται εκεί που έρχονται πρέπει να ε, είναι περίπλοκες και πρέπει να γίνουν πιο, να και πιο, να γίνουν με βάση το δικαίωμα αυτό. Και τέλος για να ε, συμφωνώ, ε, συμφωνώ με την εισήγηση και την έκθεση στο θέμα της αναβάθμισης και της διεύρυνσης των δικαιωμάτων των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες. Εκεί είμαστε σύμφωνοι, αν μπορούμε να το ενισχύσουμε περισσότερο. Στάθηκα περισσότερο σε θέματα που είτε δεν ήταν ε, ισχυρά ενισχυμένα στην έκθεση είτε θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν γιατί κατά τη γνώμη μου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η έκθεση και πρέπει να κουμπάει στη σημερινή πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ιδιαίτερος καλωσορίζω την έκθεση του κυρίου Σαλαβράκου. Είμαι δε ότι οι τροπολογίες τις οποίες θα υποβάλουν οι ε, συνάδελφοί μας θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την έκθεση. Ε, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την σύνθεση του Ευρωπαϊκού έτους, ε, του έτους για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια Ωστόσο, θα ήθελα να ζητήσω από το Προεδρείο της Επιτροπής μας να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο όταν ε, θα συζητήσουμε την έκθεση πριν την ψηφοφορία να ε, καλέσουμε είτε την Επίτροπο Ρέτινγκ είτε τον Επίτροπο Σεύκοβιτς έτσι ώστε να συζητήσουμε μαζί τους ε, το περιεχόμενο της έκθεσης. Να μην είναι απλώς άλλο ένα κείμενο, άλλη μια συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν την ολοκλήρωση της ε, τωρινής θητείας. Είναι ένα σημαντικότατο κληροδότημα το οποίο θα περάσουμε στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο επόμενο Συμβούλιο, στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι πολλά από τα προβλήματα τα οποία αναφέρονται στην ε, έκθεση, καθώς επίσης και άλλα που ανέφεραν άλλοι συνάδελφοι, θα πρέπει ορθώς να αντιμετωπιστούν στο μέλλον. Κάθε μέρα τα συζητάμε αυτά. Γιατί χάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοπιστία στα μάτια των πολιτών, γιατί φοβόμαστε ότι η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι χαμηλή, γιατί είναι πάντα η συμμετοχή στις εκλογές ε, χαμηλή. Ε, αυτά είναι τα προβλήματα. Επομένως, καλό θα ήταν να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί να δούμε ποια είναι τα προβλήματα αυτά, προβλήματα για τα οποία χρειάζεται σοβαρή συζήτηση στο μέλλον στα πλαίσια του Συμβουλίου. Προβλήματα τα οποία θα συζητηθούν και στη διάρκεια των, Ευρωπαίων εκλογών, των ευρωπαϊκών εκλογών έτσι ώστε να μην δώσουμε περιθώριο στους ε, ε, λαϊκιστές ε, να μιλάνε να δώσουμε μια πραγματική φωνή στους Ευρωπαίους πολίτες και να προσπαθήσουμε να υπεραμεινθούμε των δικαιωμάτων τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια καλή συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα. Τι θα κάνουμε δηλαδή, τι μέλη γενέστε. Γιατί αυτό είναι ακριβώς όπως έλεγα το κληροδότημά μας για την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Και στη σημερινή Ευρώπη των 28 ε, χωρών ε, μελών ήδη, ήδη υπάρχουν και κάποιοι Ευρωπαίοι πολίτες δεύτερης κατηγορίας ε, που αντιμετωπίζονται με κακό τρόπο. Ξέρουμε τι έγινε με τη συνθήκη Σέγγεν για τη Βουλγαρία, για τη Ρουμανία και άλλες περιπτώσεις όμως. Εάν θέλουμε μια πραγματική, ένα πραγματικό ε, ενωτικό μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει τα του οίκου μας πρώτα να ε, τακτοποιήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία τα οποία προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τα οποία προβλέπει η Συνθήκη Λειτουργίας και που θα πρέπει να ισχύσουν για όλους τους πολίτες, για όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχαίρω τον εισηγητή, είμαι δε πεπισμένος ότι αυτή η έκθεση θα είναι μια σημαντική συμβολή της Επιτροπής μας εδώ στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ σε όλους. Κυρίως δε ευχαριστώ τον συνάδελφο Σαλαβράκο, στον οποίο θα ξαναδώσω το λόγο έτσι ώστε να κάνει τα τελικά του συμπεράσματα ε, και στο πέρας αυτής της συζητήσεως. Ε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ε, και, και τοποθετήκαν πάνω στην έκθεση. Ε, είχα πάντα την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε μια φάση ρομαντισμού μπήκε σε μια φάση ενθουσιασμού, τώρα είμαστε σε μια φάση ρεαλισμού και προβληματισμού. Σεβόμενος αυτά τα πράγματα, προσπάθησα η έκθεσή μου να είναι κοινώ αποδεκτή από όλες τις πολιτικές ομάδες. Και παράλληλα εγνωστοποίησα προς όλους τους συναδέλφους ότι θα δεκτώ δικές τους τροπολογίες για συμπλήρωση ε, διότι θεωρώ ότι έργο του εισηγητού είναι να συνθέτει και δεν είναι να δημιουργεί εντάσεις προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Ειλικρινώς ε, ε, σας λέγω ότι στο πρώτο σχέδιο είχα περιλάβει το θέμα των μη πολιτών της Εστονίας. Είχα περιλάβει το θέμα των Ούγγρων της Σλοβακίας. Αλλά θέλησα να δώσω ένα πνεύμα στην έκθεση ε, ώστε να μην προσωποποιήσουμε σε κοινωνικές ομάδες ή σε αντιθέσεις με κράτη-μέλη διότι θα είχαμε αμέσως το σπέρμα η έκθεση αυτή να μείνει καινογράμμα. Πρέπει να περάσουμε γενικές αρχές, πιστεύω, οι οποίες να είναι ανώδυνες, να μην προσβάλλουν κανένα κράτο μέλος, αλλά να του δίνουν το έναυσμα να προχωρήσει εκείνο στις δικές του ενέργειες ούτως ώστε να έχουμε τον πολίτη της Ευρώπης διότι η νομική έννοια του πολίτου της Ευρώπης, του Ευρωπαίου πολίτη δεν υπάρχει. Η έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας είναι ιδεατή διότι όπως είπαμε η ηθαγένεια αποδίδεται βάσει της αρχής επικουρικότητας από τα κράτη-μέλη και βάσει της Ιθαγένειας εκδίδεται ένα διαβατήριο, ευρωπαϊκό <laughs> διαβατήριο δεν υπάρχει. Είναι μια σκέψη του μέλλοντος, ίσως την καλλιεργούμε με καλό τρόπο, αλλά στην παρούσα φάση στην οποία μιλάμε πρέπει να δούμε το θέμα ότι είναι πάλι στην φάση την ρομαντική, ξαναγυρίσαμε δηλαδή σε μια πιο παλιά φάση και δεν είναι στη φάση την νομική. Ε, δεν θέλω να κουράσω τους συναδέλφους, θα δεχθώ τροπολογίες και πιστεύω ότι θα βρούμε έναν τρόπο να είναι και ρεαλιστική η έκθεση και να φέρει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε και τα οποία επισήμανε και ο φίλος μου ο Βίκτορ. Ε, ευχαριστώ και πάλι για τις παρατηρήσεις του συναδέλφου. Ευχαριστώ τον κύριο Σαλαβράκο. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 16η Δεκεμβρίου. Και στις 21 Ιανουαρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και θα περάσουμε στην τελική ψηφοφορία την 10η και 11η Φεβρουαρίου στην Επιτροπή μας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Θα διακόψουμε τώρα για 10 λεπτά. Γιατί χθε αποφασίσαμε να ακυρωθεί ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Δεν κατέστη δυνατόν να έρθουν νωρίτερα τα θέματα προς συζήτηση γιατί δεν έχουμε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και αναφέροντες. Είμαστε υποχρεωμένοι για λεπτό να διακόψουμε. Θα επανέλθουμε με το σημείο 17.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 Mr. to start. Λοιπόν, ε, ξαναρχίζουμε. Παρακαλώ, καθίστε. Συνεχίζουμε λοιπόν τις εργασίες της Επιτροπής μας. Συνεχίζουμε με το σημείο 17 1441 του 12. Διντιέ Μαλέ, Γάλλος πολίτης, για τα προβλήματα που δημιουργούνται από ένα κέντρο αποβλήτων. Εκπροσωπώντας τον αναφέροντα θα πάρει το λόγο Jean-Claude Μπεκιγιόν. Έχει πέντε λεπτά για να μας παρουσιάσει το περιεχόμενο της αναφοράς του. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Bois Ρουά είναι μια αξιοσημείωτη φυσική περιοχή ε, όπου φύονται σπάνια φυτά ε, όπως αυτά του κώδικα Natura 2023-31 και επίσης ε, προστατευόμενα είδη όπως είναι το Καπριμούλγκους Ευρωπαίους καθώς επίσης και το ντεντροκόπους μέντιους ή πικ καθώς επίσης και ο ντριόκοπους μάρσιους είναι δύο είδη δριοκολάπτου αλλά κυρίως το Bois du Roi, ε, το δάσος αυτό, ε, είναι ένα μεγάλο, ε, ένας μεγάλος βιολογικός χώρος, ο οποίος συνδέει τις δασόδεις περιοχές της Βόρειας Παρισινής Κοιλάδας με αυτές των Αρδενών. Πρόκειται για ένα σύνολο το οποίο φέρει το όνομα Φορέ Πικάρντ, δάση της Πικαρδίας. Είναι το 221 2005 βάσει της οδηγίας 74 409 ΕΟΚ ένα ε, κέντρο αποβλήτων, πλατφόρμα σύνθλιψης σκυροδέματος, καθώς επίσης και επεξεργασίας μολυσμένων εδαφών ε, πρόκειται να δημιουργηθεί στο κέντρο, στην καρδιά αυτής της φυσικής περιοχής. Ο ιδιοκτήτης του Μπουάντου Ροά ε, κατάφερε να επιτύχει παράκαμψη των αμμοδών αυτών περιοχών έτσι που αναφέρονται στο Natura 2000. Ε, μία δημόσια έρευνα ξεκίνησε ε, πρόσφατα ε, έτσι ώστε να δημιουργηθούν δύο δρόμοι που θα περνούν αυτήν την περιοχή Natura 2000 και έτσι ώστε να φτάνουν, να γίνουν δηλαδή οδοί οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα σε 325.000 τόνους οικοδομικά απόβλητα να φτάνουν μέχρι την τελική εγκατάσταση. Τουλάχιστον δηλαδή 200 φορτηγά την ημέρα θα περνούν από αυτήν την περιοχή Natura 2000. Θεωρούμε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι συμβατό με, την, ε, ε, με τη διατήρηση των, ε, και την προστασία αυτών των προστατευόμενων πτηνών ε, για τα οποία δημιουργήθηκε η περιοχή Natura 2000 αλλά κυρίως θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό ε, δεν θα υπάρξει πλέον η βιολογική σύνδεση η οποία ε, υπάρχει πλέον ανάμεσα στο δάσος του Ερμενομβίλη και το δάσος του Ρέτσε. Μία επιστημονική μελέτη έγινε το 2012 από, μια, από έναν οργανισμό αναγνωρισμένο για την τεχνογνωσία του ε, πρόκειται για το AMBE ε, μελέτη η οποία επιβεβαιώνει ότι και το πέρασμα από το Bois du Roi ε, μεγάλων πτηνών καθώς επίσης και άλλων ειδών όπως είναι τα αγριογούρουνα και τα λοιπά δεν θα έχουν πλέον όλα αυτά τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας δυνατότητα επιβίωσης ή περάσματος. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή ε, ενεργοποιεί το άρθρο 10 της Οδηγίας 92-43 ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 στα πλαίσια αυτών των, ε, εργασιών της ε, για τις πράσινες και μπλε διασυνδέσεις, τραμ, βέρτε, μπλε. Παρόλα αυτά, τούτο εδώ το, το πρόγραμμα για την δημιουργία βιο, βιομηχανικού χώρου εξακολουθεί να περνάει τις διάφορες διοικητικές αποφάσει και να κοντεύει στην υλοποίησή του. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη δική σα Επιτροπή ε, όσον αφορά ε, την ελληπή εφαρμογή του άρθρου 10, παράγραφο 2, του άρθρου 18 τη Οδηγία 92 κάθε 43 κάθετο ΕΟΚ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τζαμπρίκη. Δεν έχουμε εμείς λάβει ακόμα απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το θέμα αυτό. Επομένως θα μας διαφωτίσει φαντάζομαι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Στην ουσία, ε, πάντοτε είναι αμφιλεγόμενες και δημιουργούν ε, προβληματισμούς ε, και διαφωνίες με, το, με τους περιοίκους τέτοιου είδους προγράμματα. Λαμβάνονται πάντως όλες οι πρόνοιες έτσι ώστε να γίνεται ανάλυση, αναπερίπτωση για να καλύπτονται όλες οι πλευρές ε, του πράγματος ε, και κυρίως όταν πρόκειται για δημιουργία χωματερής ε, βεβαίως λαμβάνονται υπόψη και μελετώνται από τις αρμόδιες αρχές των, κράτων μελών, των κρατών μελών συγγνώμη, όλα τα στοιχεία ε, ε, δυστυχώς όμως όποιες προσπάθειες και αν γίνονται ε, χρειάζονται οπωσδήποτε και κάποια αντισταθμιστικά μέτρα σε περίπτωση που περάσει το σχέδιο. Βεβαίως εάν δοθεί η άδεια σε παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να αναλάβει νομική δράση. Όσον αφορά την προκείμενη περίπτωση δεν υπάρχει ε, καμία απόφαση που να έχει ληφθεί όσον αφορά ε, αυτήν την ε, χωματερή. Υπήρξε η μελέτη αντικτύπου, περιβαλλοντικού αντικτύπου και στη διάρκεια αυτής θα ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία. Ωστόσο, ξαναλέω ότι άδεια δεν έχει δοθεί ακόμη και επομένως δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε διαδικασία επί ε, Εφόσον λάβουμε οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία και εφόσον τα στοιχεία αυτά αποδείξουν ότι υπάρχει παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας, οπωσδήποτε θα αναλυφθούν, ε, θα αναλυφθεί απαραίτητη νομική ε, δράση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ιτουργκάης. Ευχαριστώ. Κανονικά θα ήθελα να μεταφέρω αυτά τα οποία θα ήθελε να πει ο κύριος Μπουλάν που δεν μπορεί να είναι εδώ και θα διαβάσω ε, το σημείωμα το οποίο μου έδωσε στα γαλλικά. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να χαιρετήσω την άφηξη του εκπροσώπου του τοπικού συλλόγου. Είχα ζητήσει να υπάρξει κατεπίγουσα αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αναφοράς και την προηγούμενη εβδομάδα έμαθα ότι ήταν στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας σήμερα, αλλά εγώ δυστυχώς είμαι στην Αιθιοπία για τις ε, εργασίες των ΑΚΕ. Ε, λυπάμαι που δεν ενημερώθηκα νωρίτερα άλλωστε για την εξέταση της συγκεκριμένης αναφοράς. Παρουσιάζει ένα θέμα που ε, ενέχει κινδύνους για το τοπικό περιβάλλον και για την προστασία του περιβάλλοντος ε, στην περιοχή του Βαλουά. Οι εργασίες υποτίθεται θα ξεκινήσουν το 2014 και αυτό δημιουργεί κινδύνους και γι' αυτό ασχολούμεθα με το θέμα μέσω του μη σεβασμού των ευρωπαϊκών οδηγιών. Νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα ε, δεν τα είχα υπόψη μου πριν κάνω την δική μου παρουσίαση πριν λίγο καιρό γύρω από το θέμα και στην ουσία δημιουργείται μία χωματερή στο εσωτερικό του δάσους παραβιάζοντας ε, την περιοχή ακριβώς δίπλα από το Natura 2000. Βέβαια η μεταφορά σιδηροδρομικά ακυρώθηκε, εγκαταλείφθηκε και τώρα δεκάδες φορτηγά μεγάλα ε, σε ημερήσια βάση θα διασχίζουν την περιοχή. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ε, είναι απαραίτητη έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανεξετάσουμε το σύνολο των στοιχείων αυτού του σχεδίου μιας εταιρεία η οποία υποτίθεται ότι θα προτείνει και αντισταθμίσματα περιβαλλοντικά. Περιμένω λοιπόν κάποια επίσημη δήλωση και λυπάμαι για την έλλειψη τεκμηρίων. Ίσως αυτό να μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε σωστά το πρόβλημα και να ενημερώσουμε τους εμπλεκομένους. Ανεξαρτήτως της θέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητώ η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει επίσημα έγγραφα σχετικά με το σχέδιο το οποίο θα εξεταστεί σε περιβαλλοντικό επίπεδο και θα γίνει αντικείμενο περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων η σιδηροδρομική εταιρεία της Γαλλίας που είναι υπεύθυνη προτείνει πάντα την εκμετάλλευση των σιδηροδρομικών γραμμών και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Είναι κάτι το οποίο θίγει επίσης σαφώς και τον λεγόμενο ε, βιοδιάδρομο της περιοχής και σε επίπεδο πανίδας και σε επίπεδο χλωρίδας. Επαναλαμβάνω λέει ο μιλητής, εγώ θέλω να κρατήσουμε την αναφορά αυτή ανοιχτή. Ευχαριστώ κύριος Γιάρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τον συνάδελφο Μπουλάν. Το πρόβλημα είναι γενικό και το αντιμετωπίζουμε διαρκώς στην Επιτροπή Αναφορών. Οι χώρες μέλη μιλούν με διπλή γλώσσα. Αφενός οριοθετούν περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, φυσικού, φυσικού κάλους κλπ. Αφετέρου όταν υπάρχουν οικοδομικά συμφέροντα τις παραβιάζουν. Το πρόβλημα που βλέπουμε ξανά και ξανά είναι ότι η Κομισιόν καλόπιστα θεωρεί ότι εφόσον απλώς βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού και δεν έχει γίνει τίποτε ακόμα, θεωρούμε ότι οι χώρες μέλη θα τηρήσουν την κείμενη νομοθεσία. Στην πράξη όμως διαπιστώνουμε συχνά ότι οι χώρες μέλη προχωρούν στην δημιουργία τετελεσμένων. Αυτή τη στιγμή έχει ήδη δημιουργηθεί το συγκεκριμένο έργο, αρχίζουν και σκέπτονται πλέον μόνο για αποζημιώσεις. Δηλαδή στην ουσία συγχωροχάρτια έχουμε πολλές αναφορές δει στην ίδια κατεύθυνση και πρέπει να λεχθεί καθαρά στις χώρες μέλη ότι εφόσον έχουν οριοθετηθεί περιοχές ιδιαίτερης προστασίας οφείλουν να τηρούν τα σχετικά μέτρα και ιδίω για ε, χώρους απόθεσης απορριμμάτων αυτό είναι στην ουσία συζήτηση του προηγούμενου αιώνα θα πρέπει στην πραγματικότητα να αγωνιστούμε για να μην χρειάζεται καν να υπάρχουν χωματερές διότι η φύση από μόνη της ανακυκλώνει τα πάντα. Ο άνθρωπος ως κορονίδα της δημιουργίας θα πρέπει πρωτίστως να ανακυκλώνει. Δεύτερο, πρέπει να ζητήσω από την Κομισιόν να ζητήσει πληροφορίες από τη Γαλλική Δημοκρατία και τρίτο, να μην επιτρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα σε περιοχές προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και να καταλήγουμε σε τελεσμένα γεγονότα. Άρα, να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες της Κομισιόν και να επανέλθει να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάρ. Δεν ζητά κάποιος άλλος το λόγο, επομένως θα ξαναδώσω ε, τον λόγο στον εκπρόσωπο του ε, αναφέροντος ε, για απάντηση. Παρακαλώ. Θα ήθελα απλώς να προσθέσω μια διευκρίνηση. Όταν ε, η σιδηροδρομική γραμμή του ΤΖΒ μεταξύ Παρισιού και Βρυξέλλες ε, ε, δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε ταυτόχρονα και ένα πέρασμα πανίδος. Αυτό το πέρασμα ήταν 80 είχε φάρδος 80 μέτρα. Ένα Το μεγαλύτερο πέρασμα στη Γαλλία, αλλά ίσως και ένα από τα μεγαλύτερα περάσματα, ευρύτερα περάσματα στην Ευρώπη. Ε, πρόκειται για, ε, ένα... για μια περίπτωση εδώ, σε αυτή... αυτή την οποία συζητάμε, όπου αν δεν υπάρξει τέτοιο πέρασμα θα καταστραφεί ένα μεγάλο μέρος της προστατευόμενης πανίδας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ε, βεβαίως δεν μπορεί να σταματήσει εδώ και σήμερα αυτή η αναφορά, θα παραμείνει ανοιχτή. Θα την αφήσουμε λοιπόν ανοιχτή, ευελπιστώντας ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας ε, δώσει κάποια επιπλέον ε, στοιχεία Βεβαίω αυτή η σημερινή συζήτηση ξανανοίγει ένα θέμα το οποίο επανειλημμένα μας έχει απασχολήσει. Είχαμε και γνωμοδότηση μάλιστα ε, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, όσον αφορά τον χρόνο παρέμβασης τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Ε, δηλαδή όπω ακούσαμε και σήμερα δεν μπορεί εξ ονόματος του νόμου να παρέμβει εάν δεν έχει εκδοθεί ήδη ε, η άδεια, δηλαδή εάν δεν ολοκληρωθεί η εθνική διαδικασία αδειοδότησης. Όμως αυτό προκαλεί μεγάλο προβληματισμό στους πολίτες, προβληματισμό τον οποίο συμμεριζόμαστε και εμείς άλλωστε, ε, γιατί ε, όταν πλέον ε, φτάσει η Επιτροπή στο σημείο να μπορεί να παρέμβει, ίσως είναι πάρα πολύ αργά. Και δεν μπορούμε κι εμείς πλέον να δώσουμε μια λογική και καλή απάντηση στους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, ε, τονίζομαι προς την Επιτροπή ότι θα πρέπει κάτι να γίνει, θα πρέπει να παρέμβει και εκείνη έτσι ώστε αυτές οι δυνατότητες συνεργασίας που έχουμε και αυτές οι δυνατότητες που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να απευθυνθούν στα ενωσιακά όργανα τελικά να στέφονται από επιτυχία και να είναι επικοδομητικές, επικοδομητικές συζητήσεις. Ευχαριστώ για μία ακόμα φορά τον ε, ε, αναφέροντα και περνάμε στο επόμενο σημείο. Είναι το σημείο 18. Ε, έχουμε εδώ σημαντικό αριθμό αναφορών 1194 του 2013 της κυρίας Λίδια Πανέτο έχουμε την 1574 του 2013 του Πασκουάλε Καλδέτα στην 17-13 του 2013 που έχει υποβληθεί από τον Αλφρέντο Παλόνε, μέλος της Βουλής, Μπαρτολότσι και Καζάνα, την αναφορά πάλι της κυρίας Λάουρα Παζέτη, 1856, καθώς επίσης και την 1968 του Λουίτζι Μπούκι. Έχει καταγραφεί επίσης και η 2330 τον Αντζελίλη και Αντωνιώτση Όλες οι αναφορές έχουν κοινό θέμα το σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων στην περιφέρεια του Λάτσιο τα θέματα των χωματερών καθώς επίσης και την αποκατάσταση, εξυγίανση των χωματερών που πρέπει να κλείσουν. Λοιπόν, εγώ θα δώσω το λόγο με τη σειρά ε, των αναφορών πρώτα στην κυρία Λίντια Πανέτο. Intervengo io, non so, sono l'avvocato ε, della ε, κοιτάξτε, θα ήθελα να ευχαριστήσω, λέει ο κύριος Λίντια Πανέτο, ή ο κύριος Λίντιο Πανέτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ασχολείστε με ένα θέμα τόσο σημαντικό που αφορά τις επικίνδυνες και λιγότερο επικίνδυνες κομματερές ε, που βρίσκονται πάντα στη μέση διάταξη σε όλη την Ιταλία σχεδόν, αλλά κυρίως σε την ε, περιοχή της Ρώμης. Ε, ακόμα και ε, ε, σήμερα στην Ρώμη τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί. Ακόμα σήμερα δηλαδή φτάνουν στην ουσία όλα τα απόβλητα στις χωματερές σε περιφρόνηση πλήρη και των εθνικών νομοθεσιών αλλά και της ενωσιακής νομοθεσίας έχει δημιουργηθεί μια παράδοξη κατάσταση μη εφαρμογής ε, των ε, ενωσιακών νομοθεσιών και έχει καταλήξει βεβαίως η κατάσταση να είναι εξαιρετικά επίγουσα σε βαθμό που ε, η κυβέρνηση έχει ορίσει τον Δ. Αγκοφρέντο Σωτήλε ως ειδικό επίτροπο για την διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν υπάρχει από την Ιταλική πλευρά κανένα σεβασμός της ενωσιακής νομοθεσίας με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η ήδη εξαιρετικά βεβαρημένη κατάσταση. Ε, το ζήτημα τώρα είναι να βρεθεί μια νέα τοποθεσία για μια νέα χωματερή. Η κατάσταση πλέον είναι εξαιρετικά επίγουσα ε, και ε, πρέπει να πω ότι χωρίς να έχει γίνει προηγουμένως μια μελέτη βιωσιμότητας, χωρίς να έχει γίνει καμία τεχνική διερεύνηση και χωρίς κάποιο αρμόδιο όργανο να έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα, στα γρήγορα να ε, δίνονται κάποια νέα ονόματα ε, τα οποία όπου θα δημιουργηθούν χωματερές στην ε, αντικατάσταση της θέσεως της Μαλαγκρότα. Στην ουσία δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ότι αφήνουμε την μαλαγκρότα γιατί πλέον βρίσκονται κάποιες νέες τοποθεσίες οι οποίες έχουν επιλεγεί στην ουσία έτσι, στην τύχη. Πρέπει να πω ότι ε, η περιοχή της ε, Μαλαγκρότα είναι μια τεράστια ε, περιοχή η οποία ζει στην ουσία σε συνθήκες εγκατάλειψης πλήρους και σε συνθήκες ιδιαίτερα βεβαρημένες όσον αφορά την υγειονομική κατάσταση. Πρέπει να πω ότι γίνεται μπαλάκι μεταξύ των διαφόρων φορέων, οργανισμών, υπηρεσιών των Υπουργείων. Γίνεται μπαλάκι λέω το θέμα του ποιος φταίει και βεβαίως πέρα από την ε, ε, ε, άποψη που έχει εκφράσει ο δόκτωρ Σωτήλε, σύμφωνα με την οποία βεβαίως υπάρχει παραβίαση των, της ευνοσιακής νομοθεσίας, αυτός δεν το αναγνωρίζει και στην ουσία δεν συμφωνεί με καμία από τις εναλλακτικέ λύσεις οι οποίες υποβάλλονται βάσει του κανονισμού 98 του 2008 και που πρέπει πρέπει να ισχύσουν στη Ρώμη όπως ισχύουν ε, και σε όλες τις υπόλοιπες ε, περιοχές. Πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση της Ρώμης δεν έχουμε ούτε ανακύκλωση, ε, δεν έχουμε ούτε επεξεργασία, δεν έχουμε ούτε προσπάθεια δημιουργίας ενέργειας από, τις, από τα απόβλητα. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει σαφής παραβίαση πολλών άρθρων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και ταυτόχρονα έχουμε και ιδιαίτερη, ιδιαίτερο κίνδυνο για την υγεία των ε, κατοίκων της περιοχής. Επίσης, ε, στην περίπτωση η οποία μας απασχολεί δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα αποτροπής δημιουργίας όγκου ε, σκουπιδιών πέρα από το ότι δεν υπάρχει καμία επεξεργασία. επεξεργασία. σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει ε, η ε, χρήση της ε, μαλαγκρότα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι για μία ακόμα φορά και για τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στη Φαλκονιάνα η οποία θα έπρεπε να είχε σταματήσει τη λειτουργία της ήδη από τον Αύγουστο τίποτα δεν έχει γίνει. Πρόκειται για μία εσχρή κατάσταση πραγματικά. Ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον από τον Περιφερειάρχη, στον υπεύθυνο για τα απόβλητα της Δημαρχίας, από τον ε, υπεύθυνο επίτροπο ε, της ε, περιοχής, τον κύριο Σωτήλε, ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον και επομένως η Μαλαγκρότα έγινε επίσης το ίδιο κακόφημη, ας το πούμε, με την Φαλκονιάνα. Καταλαβαίνετε ότι και τους τελευταίους μήνες έχουμε μελετήσει το θέμα και διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πρώτον, βλέπουμε ότι ήδη από το 2003 ε, ε, ε, λειτουργεί μια χωματερή η οποία δεν κάνει κανένα διαχωρισμό ανάμεσα σε επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα. Εξακολουθεί να λειτουργεί η κατάσταση αυτή και πρέπει να πούμε ότι έχει συνεχίσει τη λειτουργία της βάση και του κανόνα πανέλη που επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι δεν επιτρέπεται βάσει αυτού του νόμου του να βάλει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ, α πούμε, ε, στην στέγη του σπιτιού σου, αλλά μπορεί ωραιότατα να εξακολουθεί να λειτουργεί μια χωματερή η οποία δεν κάνει ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε ε, επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα. Επίση, ε, κοντά στο αεροδρόμιο του Τσαμπίνο, και μερικές εκατοντάδες μέτρα από κατοικημένη περιοχή δίπλα στο Divino Αμόρε, δίπλα στο ε, πάρκο του Πιάνταντίκε των ε, παλαιών ε, φυτών κτλ. Ε, δημιουργούνται τέτοιες ε, χωματερές ε, και πρέπει να πω ότι ακόμα και η, η πρόσβαση σε αυτήν την χωματερή δεν είναι καθόλου εύκολη και επομένως το πέρασμα των μεγάλων φορτηγών με πολύ μεγάλη δυσκολία γίνεται. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν πραγματικά πώς είναι δυνατόν μια τέτοια περιοχή να θεωρείται σωστή και ότι μπορεί πραγματικά να είναι εκεί ένας χώρος υγειονομική ταφής ε, που να ε, σέβεται το όνομά του. Θα πρέπει να δούμε επίσης ε, την περίπτωση της ΕΚΟΦΕΡ, δηλαδή του φορέα διαχείρισης. Η ΕΚΟΦΕΡ έχει, αποτελείται μάλλον, είναι ένας όμιλος που αποτελείται από πάρα πολλές δεκάδες επί δεκάδων ε, ε, εταιριών και στην ουσία αυτό τι, μας οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ε, να απομονωθούν οι δραστηριότητες τους και στην ουσία δεν υπάρχει καμία διαφάνεια, επομένως μηδαμινή δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας της ΕΚΟΦΕΡ από πλευράς των ε, Ευρωπαίων πολιτών και των, των Ιταλών πολιτών. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η διαπλοκή εδώ με τη μαφία ε, είναι πάρα πολύ εύκολη. Βεβαίως έχει αποτελέσει αντικείμενο και μια σειρά ερωτημάτων στην Ιταλική Βουλή. Επίσης έχουμε φτάσει επανειλημμένα στα δικαστήρια για τα οποία, τα οποία έχουν λάβει αποφάσεις για, από φαινόμενα ότι πραγματικά ε, υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας, ότι πραγματικά υπάρχει υπάρχει ε, μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας ε, λόγω της μόλυνσης που προκύπτει από αυτόν τον τρόπο διαχείρισης ε, των αποβλήτων. Η δημόσια διοίκηση της Ιταλίας θα πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της. Θα πρέπει κάτι να γίνει για όλα αυτά. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί μακρηγόρησα και να σας ευχαριστήσω που κρατάτε αυτή την αναφορά ανοιχτή. Ευχαριστούμε πολύ. Να χαιρετήσω την αντιπροσωπεία της Ιρλανδικής Βουλής που ασχολείται με τα δικά μας θέματα. Είναι χαρά μας που σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ και θα ακούσουμε αργότερα και μία παρέμβαση από τη δική σας πλευρά κατά τη διάρκεια της πρωινής πάντα συνεδρίασης. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σήμερα. Θα περάσουμε στον επόμενο πολίτη αναφέροντα Ο κύριος Καλτσέτα έχει το λόγο για λίγα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους εκπροσώπους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διαχείριση των αποβλήτων στο Λάτιο ε, δεν σέβεται τους κανόνες ούτε τους Ιταλικούς ούτε τους Ευρωπαϊκούς. Αναφέρομαι εδώ στην Οδηγία 2008 την απόφαση του Συμβουλίου του 2008 πάλι, που προτείνει την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση ε, και όχι ε, την καύση ή την αποθήκευση των αποβλήτων. Υπάρχουν ε, άλλες εναλλακτικές λύσεις περισσότερο αποδεκτές. Έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις, έχουμε οδηγηθεί στην περιοχή της επαρχίας της Ρώμης σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Στην περιοχή της Φαλκονιάνα αποφασίστηκε να γίνει ακριβώς η αποθήκευση των αποβλήτων της πρωτεύουσας. Η απόφαση ελήφθη το 2013 τον Αύγουστο τη νύχτα σε μια συνάντηση όπου συμμετείχε ο Αντρέο Ορλάντο, Υπουργό Οικονομικών, όπως επίσης και ο Ινιάτσιο Μαρίνο, δήμαρχος της Ρώμης, και ο κύριος ζητήθηκε από τον Σωτήλε να επαληθευθούν σε επίπεδο επιμελητίας οι δυνατότητες της συγκεκριμένη αυτής περιοχής. Υπήρξαν διαμαρτυρίες από τις δημοτικές αρχές των γειτονικών χωριών και οικισμών Ζητήθηκε και από το Εθνικό Κοινοβούλιο να λάβει θέση, κατετέθησαν αρκετά διαβήματα, υπήρξαν αρκετά διαβήματα των τοπικών αρχών. Όλοι οι υπουργοί οι οποίοι αναφέρονται ε, στις, στα διαβήματα αυτά έχουν επαναλάβει ότι ε, τους δόθηκαν γνωμοδοτήσεις από πλευράς του Επιτρόπου Σωτήλη. Ο υπουργό Μοάβερο είπε ότι ποτέ δεν ζητήθηκε ουσιαστικά η γνώμη του. Ο υπουργό Εσωτερικών είπε επίσης ότι ε, δεν του ζητήθηκε επίσης από τον Επίτροπο ό,τι λέει η εξέταση ε, των ε, ιδιωτήτων αν θέλετε και των χαρακτηριστικών της επιχείρησης η οποία είναι υπεύθυνη για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ε, και σε επίπεδο περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και η ε, συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται από, τις, από τους ισχύοντες κανονισμούς στην περιοχή. Δεν ζητήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ε, ε, μελέτη για τις ε, επιπτώσεις στον τομέα της υγείας και ο Υπουργός Τζιρόλαμο του τομέα της Γεωργίας είπε ότι δεν ζητήθηκε ούτε η δική του άποψη. Τελικά ο Υπουργός Ορλάντο, αυτός ο οποίος παρέπεψε το θέμα στον Ειδικό Επίτροπο, είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε την δυνατότητα να εξετάσει τις δηλώσεις Άγια και που έγιναν από τους... Όλες αυτές οι δηλώσεις έγιναν επαναλαμβάνω από τους υπουργούς στο εσωτερικό της Ιταλικής Εθνοσυνέλευσης. Ο συγκεκριμένος Επίτροπος Περιβάλλοντος είπε ότι για τις δυσκολίες ε, επικοινωνίας δεν υπάρχει δυνατότητα. Στην Βία Αρντεατίνα υπάρχει μια λωρίδα για τα φορτηγά την οποία βέβαια δεν σέβεται κανείς ε, και θα μπορούσαν και τα φορτηγά που θα μεταφέρουν τα απορρίμματα να μην σέβονται και αυτά τον συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Η κατάσταση λοιπόν είναι απαράδεκτη. Οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους πολίτες και γι' αυτό ακριβώς καταθέσαμε την αναφορά ζητώντας την παρέμβασή σας έτσι ώστε να ελέγξετε το σεβασμό των ισχυουσών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης ε, των αστικών απορριμμάτων. Ε, να αξιολογηθεί εκ νέου η περιοχή της Φαλκονιάνα και να δοθούν εγγυήσεις στους πολίτες οι οποίοι εμπλέκονται για την σωστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Ζητάμε λοιπόν από τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής να στηρίξουν τη συγκεκριμένη αναφορά έτσι ώστε η αδειοδότηση να δοθεί ελέγχοντας όμως πλήρως τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Λάουρα Παζέτη. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής και με την ε, δικιά μου ε, αναφορά ε, θα θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε την πολύ άσχημη κατάσταση και η οποία κάθε μέρα χειροτερεύει στην περίπτωση της Φαλκονιάνα μετά από το κλείσιμο της Μαλαγκρότα πολίτες ε, συζητούν διαρκώς το θέμα ε, ε, και φοβούνται ότι οπωσδήποτε σε περίπτωση που ανοίξει η χωματερή της Φαλκονιάνα θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή. Ε, γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που ανοίξει ε, η, Φαλκονιάνα οπωσδήποτε θα υπάρχει παραβίαση της υφιστάμενης ε, ενωσιακής νομοθεσίας και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα κυρίως διότι στις γειτονικέ περιοχές υπάρχει γεωργική καλλιέργεια συγκεκριμένων ειδών ονομασίας, προστατευόμενης ονομασίας Επίση, Επίσης, να μην λησμονούμε ότι η περιοχή ε, παρουσιάζει υψηλό βαθμό σεισμικού κινδύνου. Η αδειοδότηση θα πρέπει να γίνει μονάχα ε, και εφόσον ξεπεραστούν τα προβλεπόμενα από ε, περιβαλλοντικούς κανονισμούς, όπως ας πούμε ο κανονισμός Bondi ε, που ισχύει στην Ιταλία. Η ιδιαίτερα μεγάλη περατότητα των πετρωμάτων του υπεδάφους της συγκεκριμένη περιοχής και το πέρασμα από πολύ κοντά του ποταμού Τίβερη στην περιοχή της Βαλκονιάνου ε, δημιουργούν επιπλέον προβλήματα. Θα πρέπει επομένως να γίνουν πολύ προσεκτικά οι μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου ε, γιατί ε, βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση που δοθεί η αδειοδότηση θα δημιουργηθούν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία θα είναι οικολογικά, περιβαλλοντικά αλλά θα αφορούν και την υγεία του πληθυσμού. Επίσης ε, θα ήθελα να πω ότι ε, η πρόσβαση ε, της, στις περιφέρειες, τις γειτονικές της Φαλκονιάνα ήδη είναι προβληματική λόγω της εγκύτητας της Βία Λαουρεντίνα και βεβαίως θα επιβερυνθεί περαιτέρω και με ιδιαίτερα άσχημο τρόπο εάν αρχίσει και η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στην ίδια περιοχή το άρθρο 32 του, ε, ε, του Ιταλικού Συντάγματος ε, δίνει την δυνατότητα προστασίας, προβλέπει μάλλον την προστασία της υγείας των πολιτών και στην προκείμενη περίπτωση βλέπουμε ότι θα υπάρξει παραβίαση αυτού του άρθρου. Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν ενωσιακοί κανόνες όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας σε σχέση ε, με τους χώρους ε, ταφή ε, απορριμμάτων. Να μην λησμονούμε επίσης ότι ήδη από το 2011 έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραβάση για, την, για τη Μαλαγκρότα και που βασίζεται σε χαρακτηριστικά παρόμοια με τα χαρακτηριστικά που θα έχει η χωματερή τη Φαλκονιάνα. Είτε πρόκειται για τον τρόπο μεταφοράς, είτε για τον τρόπο απόρριψη των αποβλήτων, είτε για την αποτροπή δημιουργίας αποβλήτων, την μη επεξεργασία κτλ. Όλα στοιχεία τα οποία τελικά επιβαρύνουν την δημόσια υγεία. Ε, εμείς θα θέλαμε να ε, ε, υπάρχει επεξεργασία των απορρεμάτων, πράγμα που δεν προβλέπεται στην Φαλκονιάνα. Προβλέπεται μονάχα σύνθλιψη και εν τέλει αποτέφρωση των απορριμμάτων, των απορριμμάτων συγγνώμη, χωρίς καμία προηγούμενη επεξεργασία. Η Επιτροπή η οποία αναφέρθηκε, η οποία ασχολήθηκε μάλλον με την μελέτη του θέματος ε, ε, ε, δεν έχει δώσει καμία δεν έχει δώσει κανένα θετικό στοιχείο όσον αφορά την Φαλκονιάνα. Θα πρέπει οπωσδήποτε η Ιταλική κυβέρνηση να προβλέψει χώρους απόρριψης και επεξεργασία των απορριμμάτων έτσι όπως προβλέπονται και από την Ενωσιακή νομοθεσία. Ε, θα, στην ε, Μαλαγκρότα είδαμε τι έχει γίνει. Παρόμοια κατάσταση θα προκύψει και στην ε, Φαλκονιάνα σε περίπτωση που δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Επίσης στην Φαλκονιάνα δεν έχουν ακολουθηθεί οι σωστές διαδικασίες όσον αφορά την αδειοδότηση. Έχουμε πολλά προβλήματα όσον αφορά την απόρριψη ε, ακόμα και επικίνδυνων μολυσμένων αποβλήτων, νοσοκομιακών αποβλήτων κλπ. Ε, αυτό θα σημαίνει ότι και τα σωματίδια της σκόνης καθώς επίσης ε, και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ξέρουμε ότι η Ιταλική κυβέρνηση έχει ορίσει ειδικό επίτροπο για τα απόβλητα ε, ωστόσο δεν έχει προβλέψει κολεγιακές διαδικασίες όσον αφορά την λήψη των αποφάσεων. Ε, στην προκείμενη περίπτωση ε, αναρωτιέμαι και γι' αυτό ακριβώς έχω υποβάλει την αναφορά ενώπιόν σας. Αναρωτιέμαι εάν είναι δυνατόν να σταματήσει η δημιουργία της Φαλκονιάνα ή εν πάση περιπτώσει να προχωρήσει η αδειοδότηση με διαφορετικό τρόπο από ότι αυτή της Μαλαγκρότα. Να μην λησμονούμε ότι δίπλα στη Μαλαγκρότα υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, περιοχές ε, οι οποίες παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον όπως είναι το Κόλεντι Πίντε, τα Παλώμα, τα Φιούμια κτλ. Οι Ιταλικές ε, αρχές ε, θα πρέπει να σταματήσουν, ε, να, σταματήσουν τη διαδικασία δημιουργίας χώρου απόρριψης απορριμμάτων. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος και δίνω το λόγο στον επόμενο παρεμβαίνοντα. Ο κύριος Μπούκη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Αναφορών, η απαράδεκτη ιστορία στον Δήμο του Μπρατσάνο ξεκίνησε από το 1990 μετά την αποκατάσταση μιας παλαιάς χωματερής παράνομης. Θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί για τρία χρόνια το πρόβλημα των απορριμμάτων ε, με βάση την απόφαση 4509 του 90 η συγκεκριμένη χωματερή στο Κουπινόρο θα έπρεπε να παίρνει τα απορρίμματα 8 χωριών ε, γύρω. Αλλά σήμερα είναι 25 οι κοινότητες οι οποίες μεταφέρουν εκεί τα απορρίμματά τους και 4 ιδιωτικές εταιρείες. Έχει προβλεφθεί πολλές φορές να κλείσει η συγκεκριμένη χωματερή ε, έχουν ε, διαδεχθεί στην διαχείριση της χωματερής ε, πάρα πολλές εταιρείες και τα τελευταία χρόνια τη διαχειρίζεται η μια επιχείρηση του Δήμου του Μπρατσάνο. Τους επόμενους μήνες περιμένουν 20.000 τόνους που προέρχονται από τη Ρώμη, το Τσαμπίνο, το Φιουμιτσίνο και την πόλη του Βατικανού επί τη βάση ακριβώς του προγράμματος της εταιρείας Μπρατσάνο Ambiente η χωματερία αυτή θα διευρυνθεί ε, με 450.000 τετραγωνικά ε, κυβικά μέτρα θα έλεγα και με απόφαση της 16ης Οκτωβρίου του 12 η περιφέρεια του Λάτιου έδωσε θετική γνωμοδότηση και προβλέπεται ακριβώς η δημιουργία ενός βιομηχανικού κέντρου επεξεργασίας απορριμμάτων με εγκαταστάσεις TMB και παραγωγής βιοαερίου, χωρίς να ακουστεί καθόλου η άποψη των πληθυσμών που ζουν κοντά στην περιοχή της Χωματερής, σε μια ζώνη η οποία ονομάζεται ε, ΖΠΣ, δηλαδή ειδική προστασίας περιοχή και πολύ κοντά στην ε, ε, μεσαιωνική πόλη του Τσέρι και στη λίμνη του Μπρατσάνο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια συμπληρωματική αύξηση του χώρου, ιδιαίτερα μετά από το κλείσιμο της Μαλαγκρότα όπου για 30 χρόνια δεχόταν τα απορρίμματα της Ρώμης έχουμε να κάνουμε με ένα ξεπερισμένο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ υπάρχουν νέου τύπου οδηγίες και το θέμα οδηγείται σε αδιέξοδο. Πρόκειται για ένα αδιέξοδο το οποίο είχε, θα έλεγα, ανακοινωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, λόγω ακριβώς της καθυστέρησης ε, την οποία σημείωσαν όλοι οι δήμοι της περιοχής του Λατίου λόγω των διοικητικών και οικονομικών αδυναμιών των περιφερειακών εκτελεστικών αρχών. Ε, για μια ακόμη φορά λοιπόν χρειάστηκε ένα υπουργικό διάταγμα το οποίο δίδει πολλές αρμοδιότητες στον ειδικό επίτροπο ε, για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Ρώμης ο οποίος θα μπορεί επίσης να αποφασίζει για το πότε θα μεταφέρονται τα απορρίμματα της πρωτεύουσα στο Κουπινόρο. Ε, το επισκεφθήκατε αυτό στις 7 Νοεμβρίου και στην ουσία ονομάζεται η περιοχή του Κοπινόρο η Μαλαγκρότα των Φτωχών, χωρίς έλεγχο ε, εισόδου, ε, με ε, πραγματικά παρακμιακή κατάσταση, εγκαταλελειμμένες ε, εγκαταστάσεις και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η Ιταλία έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την κακή διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή του Λατίου. Α, κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος λοιπόν της Επιτροπής του Μπόργκο Σαν Μαρτίνο τη ε, της Επιτροπής εναντίον της ε, χωματερής του Τσερβέτερη ε, και με βάση την αναφορά 1968 του 2013 επί τη βάση όλων αυτών τα οποία προείπα, λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα του προβλήματος και λόγω του ότι η μοναδική αρχή που γίνεται η σεβαστή είναι ότι το προσωρινό μονιμοποιείται, δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα και υγεία αύξηση σαν παράδειγμα των καρκινικών όγκων στον πληθυσμό του Λατίου και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ρίξει φως ε, επί τη βάση της συγκεκριμένης αναφοράς. Σας ευχαριστώ πολύ που σεβαστήκατε το χρόνο. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο ο οποίος είναι ήδη ενημερωμένος για τα θέματα αυτά, αν και αντιμετωπίσαμε την αναφορά με κατεπήγοντα τρόπο. Γιατί το αντικείμενο των συγκεκριμένων αναφορών είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό θέμα γνωστό στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ελπίζουμε να λειτουργήσει σωστά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, η Κομισιόν γνωρίζει καλά την κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων στο Ρωμαϊκό Λάτσιο αλλά και γενικότερα στην Ιταλία αλλά προσπαθήσαμε για ένα διάστημα σε συνεργασία με τις Ιταλικές Αρχές να εξεύρουμε κάποια λύση για την κατάσταση νομίζουμε ακούσαμε τις αναφορές γνωρίζουμε που βρίσκεται το πρόβλημα και θεωρούμε ότι η λύση έγκυται στην έγκριση των σωστών σχεδίων διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως και αλλού στην Ευρώπη. Οι Ιταλικές αρχές το έπραξαν αυτό και στο Λάτσιο, αλλά αυτά τα σχέδια πρέπει τώρα να εφαρμοστούν όπως είναι στα χαρτιά. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την χρήση των χωματερών, αν και Σαφώς η απόψή μας είναι ότι οι χωματερές θα έπρεπε να βρίσκονται τελευταίες στην ιεραρχία και θα έπρεπε να υπάρχουν άλλα, άλλοι τρόποι διαχείρισης των απορριμμάτων. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο Λάτσιο. Παρόλα αυτά, η Κομισιόν θεωρεί ότι οι χώρες μέλη διαθέτουν περιθώριο διακριτικής ευχέρειας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε ό,τι αφορά την επιλογή των μεθόδων διαχειρίσεως των απορριμμάτων. Η χωματερή είναι μία από τις μεθόδους αυτές. Και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα βέβαια στο Λάτσιο είναι η μαλαγκρότα η οποία έκλεισε τώρα και τώρα πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων. Συμφωνούμε με τους αναφερομένους ότι θα έπρεπε να έχουν ήδη εξευρεθεί λύσεις διότι η Μαλαγκρότα δεν είναι και τίποτε το νέο και τα σχέδια για το κλείσιμό της υπήρχαν εδώ και χρόνια. Γνωρίζουμε επίσης τις ενδεχόμενες επιλογές Φαλκονιάνα και Κουπινόρο. Αυτό που είναι σημαντικό να λεχθεί ωστόσο είναι ότι η Κομισιόν μπορεί να παρέμβει μοναχά δυνάμει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας μόνο εφόσον διαθέτει ενδείξεις ότι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις απόρριψης των απορριμμάτων έχουν εγκριθεί και λειτουργούν κατά παράβαση των Ευρωπαϊκών Διατάξεων Διαχείρισης των Απορριμμάτων, Μελετών και Αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών Αντικτύπων και της σχετικής διαχείρισης. Η διαδικασία έγκρισης, ωστόσο, αδειοδότησης, είναι στα χέρια των εθνικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο όταν οι απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, για παράδειγμα επαρκής διαβούλευση του κοινού και επαρκής μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, έχουν παραβιαστεί. Τέτοια στοιχεία δεν έχουμε λάβει ακόμη. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να λάβει τέτοια. Έχουμε τώρα κάποια γνώση και των σχεδίων για την περίοδο μετά την Μαλαγκρότα στο Λάτσιο εξήγησε η Επιτροπή στις Ιταλικές Αρχές ότι όλη η εφαρμόσιμη ευρωπαϊκή νομοθεσία, οδηγία περί χώρων απορριμμάτων, χιτά δηλαδή και άλλες, πρέπει να τηρηθούν. Οι Ιταλικές Αρχές τα γνωρίζουν και περιφερειακές και εθνικές. Θα παρακολουθήσουμε τις συγκεκριμένες επιλογές τις οποίες θα προβούν για τις χωματερές και αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν στοιχεία ότι έχει παραβιαστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση. Όπως λέχθηκε ήδη, υπάρχει ήδη ανοιχτή διαδικασία για παραβίαση κατά της Ιταλίας σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων, όχι μόνο στην Μαλαγκρότα, που έκλεισε όμω τώρα, αλλά και ως ολόκληρη την περιοχή του Λάτσιο, διότι θεωρούμε ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και πριν από τη χωματερή. Αυτή η διαδικασία κρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αναμένουμε την απόφασή του. Σύντομα. Θα ολοκληρώσω το σχόλιο μου λέγοντας ότι η Κομισιόν είναι ανοιχτή να δεχθεί οποιαδήποτε ένδειξη που μπορεί να δείχνει κάποια παραβίαση αλλά θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη το γεγονό ότι ναι μεν δεν μπορούμε να παρέμβουμε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην διαδικασία για την επιλογή των χωματερών εφόσον βέβαια τηρούνται οι διατάξει τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ωστόσο αυτή η επιλογή γίνεται στο επίπεδο της χώρας μέλους είτε εθνικό είτε περιφερειακό αναλόγως με τη δική της νομοθεσία Thank So... Σας ευχαριστώ πολύ Θα αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση Πρώτα η κυρία Άουκεν. Πρόκειται για μια ιστορία σε συνέχειες. Και πολλοί από τους αναφερομένους και τους πολίτες, όχι μόνο στο Λάτσιο αλλά και στην καμπάνια, παρακολουθούν το τι συμβαίνει εδώ και εκπλήσονται που βλέπουν την Κομισιόν πάλι παράλυτη, να λέει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Παρόλο που είναι μια Διαρκή ιστορία. Καμιά φορά αντιδρά η Κομισιόν, καμιά φορά δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Όταν είχαμε πάει εκεί σε αποστολή την τελευταία φορά πέρσι, ακούσαμε συγκεκριμένα στοιχεία επιτράπη, συνεχίζεται η ίδια πραγματικότητα. Νόμιμες παράνομες χωματορές χωρίς συμμετοχή των πολιτών, χωρίς να γίνεται καμία πρόσκληση για επιλογή των απορριμμάτων, να τους ζητήσουν δηλαδή να τα ξεχωρίζουν κτλ. Άρα δηλαδή με τη δική σας στάση θα συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Και από ό,τι βλέπω η Κομισιόν γίνεται χειρότερη από ό,τι ήταν. Εμείς αναμένουμε από την Κομισιόν να αντιδρά. Όταν έρχονται οι πολίτε και μας λένε ότι οι οδηγίες δεν τηρούνται. Εμεί το βλέπουμε αυτό. Και ιδίω η οδηγία περί απορριμμάτων. Λέμε σε ορισμένου από τους αναφερομένους. Εμείς έχουμε κάνει πολλά λάθη στη Δανία και πολλές λάθο επιλογές και επενδύσεις. Εμείς τα ρίξαμε όλα στην καύση. Προσπαθούμε τώρα να βρούμε άλλους νέους τρόπους να ανακτήσουμε πόρους από τα απορρίμματα αντί για αυτή την ανόητη πολιτική της καύσης και η Ιταλία να μην επαναλάβει τα λάθη τα δικά μας να προχωρήσει ευθέως στην ανακύκλωση να φτιάξει δηλαδή μια κυκλική οικονομία διαχείρισης των αποβλήτων. Είναι όμως πραγματικά ο κόδρας του κινδύνου. Όταν ακούμε ότι η Κομισιόνα λέει ότι ήταν από την αρχή καθαρό ότι ήταν έκτακτη η κατάσταση, αλλά μετά τα βρήκε όλα νόμιμα. Και εμείς πήγαμε και είδαμε υπέροχέ τοποθεσίες κοντά στο Βεζούβιο και αλλού, που μάλιστα υπήρχαν και στρατιωτικές φρουρές με την πρόφαση «Α, είναι έκτακτη κατάσταση. Εφόσον δεχτούμε τέτοια πράγματα, εφόσον δηλαδή τα δεχθεί η Κομισιόν τα πράγματα αυτά, ξεπηδούν πολλά ερωτήματα. Εγώ έχω πολλές ερωτήσεις προς εσάς, αλλά μου φαίνεται λίγο παράλογο να σας κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις, τι θα γίνει δηλαδή με το α, με το β, με το γ μέρος, που τα είδαμε όταν είχαμε πάει εκεί, όταν ακούω από εσά τώρα ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει και ίσως έκλεισε η μαλαγκρότα καλά, αλλά δεχόμαστε να φτιαχτούν άλλες χωματερές χωρίς να ληφθεί κανένα μέτρο προφύλαξης. Θα ήθελα να ακούσω, εάν πραγματικά σκέφτεστε ότι η Κομισιόν πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή, δεν... ή ξαναρχίσει από το μηδέν. Τέλος, νομίζω ότι πρώτα-πρώτα πρέπει να ζητήσουμε σε όλες τις περιπτώσεις αυτές σε όλες τις περιπτώσεις αυτές να ζητήσουμε τη συμμετοχή των πολιτών. Αυτό το πρόβλημα σημειώθηκε στην καμπάνια, στο Λάτσιο, της Ρώμης. Αν δεν εμπλακούν οι πολίτες, ποτέ δεν θα κερδίσουμε. Και επειδή η Επιτροπή μας είναι η Επιτροπή των Πολιτών, οφείλει να επιμείνει σε αυτή τη συμμετοχή των πολιτών όπως είδαμε στην αρχή, στην Άπολη Ο είδαμε δηλαδή μια απαρχή της συμμετοχής αυτών των πολιτών, αυτή των πολιτών και επίσης να επιμείνουμε σε πλήρη διαφάνεια ώστε ο καθένας να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το τι γίνεται αντί να υπάρχουν αυτά, αυτές οι έκτακτες καταστάσεις με στρατιωτικές φρουρές κτλ όπου κανείς έχει την αίσθηση ότι πάνε εκεί να συγκαλύψουν δεν θέλω να πω εγκληματικές ενέργειες όσο είναι υπερβολικά δραματικό πάντως Κανείς δεν γνώριζε περί τίνος επρόκειτο, τουλάχιστον όσοι ήθελαν να είναι καθαροί απέναντι στην νομοθεσία. Παρακαλώ τους συναδέλφους να μην μιλούν περισσότερο από τους ίδιους τους πολίτες. Η κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους αναφέροντες. Εμείς ακούμε για μια κατάσταση κατεπήγοντος και ακριβώς ε, οι καταστάσεις ε, κατεπήγουσες ε, οδηγούν στην δημιουργία θέσεων ειδικών επιτρόπων. Το ακούσαμε και στην Άπολη, το ακούμε και για στο, στην περίπτωση του Λάτιου. Και εδώ έχουμε τον Επίτροπο Σωτήλε, τον συναντήσαμε πέρυσι κατά τη διάρκεια της αποστολής μας και ήταν σαφές ότι ο συγκεκριμένος κύριος έχει πάρα πολλές διευρυμένες αρμόδιότητες για την αντιμετώπιση αυτής της κατεπίγουσας κατάστασης σχετικά με τα απορρίμματα. Διαρωτώ με εδώ αν κάτι τέτοιο η διαδικασία αυτή είναι δημοκρατικά νόμιμη. Δεν αναφέρομαι μόνο στην οδηγία πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά έχουμε ένα έκτακτο επίτροπο να παρεμβαίνει σε τομείς όπου ο Υπουργός και το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχουν την τελική ευθύνη. Διερωτώμε λοιπόν αν κάτι τέτοιο είναι πραγματικά εφικτό σε μια δημοκρατική Ευρώπη και σε ένα δημοκρατικό σύστημα σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του καθενός. Τώρα ακούμε για έκτακτα σχέδια και ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι ε, επανέρχεται στα θέματα της διαχείρισης ε, από συγκεκριμένες μονάδες των αποβλήτων. Τα είδαμε και στην Νεάπολη της Ιταλίας Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν το τον κατεπήγοντα χαρακτήρα. Πρέπει να ξεπεράσουμε το στάδιο αυτό και πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί βλέποντας το τι χρειάζεται να γίνει πριν δημιουργηθούν τα προβλήματα αυτά στις χωματερές και πριν δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες χωματερές ή παρατηρηθούν ότι λειτουργούν. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάποιες ε, ιδιαίτερες δυσκολίες με την καύση των απορρίτων, των αποβλήτων. Ε, ξέρω ότι αυτό είναι πρόβλημα όμως και στην περιοχή της Καμπανίας ε, και στο Λάτιο. Να μου πει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως είναι δυνατόν οι πολίτες να μην είχαν καμία δυνατότητα έκφρασης. Γιατί οι πολίτες πρέπει να προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν τελευταία προσφυγή. Δεν είναι δυνατόν να κινητοποιηθούν νωρίτερα, δεν είναι δυνατόν να γίνει πιο προληπτική η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τους συναδέλφους. Συμφωνώ μαζί τους. Ωστόσο θα ήθελα να επανέλθουμε στο κεντρικό πρόβλημα που είναι ε, το θέμα της Φαλκονιάνα. Βεβαίως ε, η γενική συζήτηση για το περιβάλλον στην Ιταλία είναι ιδιαίτερη. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπατε, αλλά να μην ξεφύγουμε από το θέμα. Εγώ άκουσα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και κυρία Πρόεδρε πραγματικά εκπλήσωμαι. Ίσως καλύτερα είναι να διαβάσει κανείς τη δίκη του Κάφκα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν κατάλαβα στην ουσία αυτό που μας είπε. Ή μάλλον, να το πω καλύτερα, πολύ καλά κατάλαβα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Οι αδειοδοτήσεις που δίνει η Ιταλική κυβέρνηση, οι επιλογές που κάνει. Η συζήτηση γίνεται πάντα εκ των υστέρων και δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ε, ε, υπέβαλα και μία ερώτηση ως βουλευτής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ζήτησα από τον Επίτροπο με ε, φάκελο για το περιβάλλον ορισμένα πράγματα. Πρώτον, επαλήθευση των ε, ε, προϋποθέσεων για την δημιουργία της Φαλκονιάνα. Δεύτερον, έλεγχο όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών. Τρία, την επαλήθευση των ε, διαδικασιών που ακολούθησε η περιφέρεια του Λάτσιο ε, όσον αφορά την συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κοιτάξτε αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς δεν θέλουμε γραφειοκρατική Ευρώπη. Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία θα είναι πάντοτε παρούσα. Η στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρώπη. Και τι μου απήντησε ο Επίτροπος, και αυτό είπε προηγουμένως για τον Κάφκα. Ο, ο κύριος Ποτόσνικ λοιπόν μου απήντησε στα πλαίσια της διαδικασίας υπεπαράβαση τάδε τάδε ε, όσον αφορά την ε, ε, μαλαγκρότα. Αναφέρεται δηλαδή στην, στον χώρο απόρριψης της μαλαγκρότα. Μπορώ να σας πω ότι η περιφέρεια του Λάτσιο δεν έχει τις απαραίτητες συνθήκες έτσι ώστε να κάνει διαχωρισμό και επεξεργασία των απορριμμάτων. Θα ληφθούν υπόψη ή θα ληφθούν υπόψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε και... Δηλαδή δεν χρειάζεται να να περιμένουμε να χτιστεί η νέα μονάδα έτσι ώστε να παρεύουμε. Όμως εδώ η διαδικασία είναι καυκική. Ε, επίσης συνεχίζει η απάντηση και μου λέει ναι δεν γίνονται σεβαστές ε, οι προϋποθέσεις. Άρα τι μου λένε δηλαδή ότι στην, περιοχή του Λάτσιο υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά ε, τα σκουπίδια. Δηλαδή είτε το δεχόμαστε είτε, είτε θα γίνουμε όλοι παλαβοί. Θα πρέπει να κλειστούμε σε φρονοκομείο. Δηλαδή, από τη μία μα λένε ναι, υπάρχει Ευρώπη, ναι, υπάρχουν κανόνε. Από την άλλη μα λένε ναι, οι κανόνε δεν έχουν γίνει σεβαστοί. Αλλά εμεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε παρόλα αυτά τώρα. Τι θα κάνουμε δηλαδή εδώ. Και ξέρετε, νομίζω ότι ε, ε, ε, λέει ακόμα ο Επίτροπος, ορισμένα ε, χώροι, ε, στο, ορισμένες χωματερές στο Λάτσιο ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουν σε επεξεργασία των απορριμμάτων πριν την απόρριψή τους στην χωματερή, γιατί διαφορετικά υπάρχει παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας 2008 κλπ, κλπ η οποία αναφέρεται στην επεξεργασία των απορριμμάτων. Τι να πω δηλαδή, μπορούμε να περιμένουμε πλέον να χτιστούν αυτές οι μονάδες και μετά ε, να παρέμβουμε και μετά να, κάνουμε, να, να πάρουμε ποιον, τον κυβερνήτη, την περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον, τον ε, υπουργό ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και λέει ότι ναι θα δοθεί η άδεια εάν, ε, αναφέρομαι τώρα πάντα στην απάντηση που μου έδωσε ο κ. Ποτόρνικ, ε, ε, ε, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα εάν δεν γίνει σεβαστή η ενωσιακή νομοθεσία. Μα τι λέει τώρα, αφού έτσι κι αλλιώ ξέρουμε ότι δεν έχει γίνει σεβαστή η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Λέει το ίδιο, το αντίθετό του, φάσκη αντιφάσκη. Πρώτα μας λέει ότι δεν υπάρχει ε, η μονάδα, μετά μας λέει ότι όταν θα γίνει ε, τότε θα πάρουμε μέτρα, μετά μας λέει ότι έχει γίνει άρα δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα. Κάφκα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ε, δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ένα ολόκληρο βιβλίο για το, για το θέμα του Λάτσιο. Η κυρία Αντζελίλη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω πάρει πάρα πολύ τεκμηρίωση εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω φυσικά τους συναδέλφους Παλώνε και Αντωνιώτσι, με τους οποίους πράγματι αποτελούμε μια ισχυρή ομάδα. Πέρα από τον αναφερόμενο και τους υπόλοιπους αναφερομένους, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους παρόντες οι οποίοι είναι εδώ και δεν ομιλούν. Αλλά εγώ θα είμαι η δοκή τους φωνή σαν παράδειγμα του Αρμάντο Τολτινέλη, Δημοτικού Συμβούλου του, α, της περιοχής, του Αλεσάντο Γκράντο, της Φρανκασούτο, του Στεφανέλη, ε, του Περιφερειακού Πάρκου του Μπρατσάνου, της Επιτροπής ε, Εναντίον των Αποβλήτων στο Μπρατσάνο, της Άννα Ορτσίνη, ε, τους Δημοτικούς Συμβούλους Μπονέλη και Ντενάπολη, τους εκπροσώπους των ε, συγκεκριμένων συλλόγων για την προστασία του περιβάλλοντος κτλ. Σταματώ εδώ στην απαρίθμηση όλων αυτών που δεν μπόρεσα να μιλήσω, αλλά ήθελα να πω ότι έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό επανειλημμένα. Πέρυσι είχαμε κάνει και ένα έκτακτο ταξίδι, μια μορφή επίσκεψης ερευνητικής στα θέματα που αφορούν στις περιοχές ε, μάλλον που ε, ασχολούνται με την επεξεργασία των απορριμμάτων της Ρώμης. Και αυτό το είπε πολύ σωστά ο συνάδελφος Παλώνε. Έχει παραπεμφθεί η Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εδώ και δεκαετίες περίπου ε, λειτουργεί το σύστημα της επιτροπίας, μια επιτροπία η οποία τις, τα τελευταίες, ε, τους τελευταίους δύο χρόνους ε, έχει βρει κάποιες επιπλέον περιοχές ε, για χωματερές και απαριθμη τις χωματερές αυτές η κυρία Αντζελίλη. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Από προσωρινή χωματερή σε προσωρινή χωματερή δεν βρίσκουμε ποτέ μόνιμη χωματερή και συνεχίζεται ο κατεπήγον χαρακτήρας της αντιμετώπισης του προβλήματος, παραβιάζοντας φυσικά τους κοινοτικούς κανόνες, μη σεβόμενοι τα δικαιώματα των πολιτών, παραβιάζοντας τα χωροτεκτικά σχέδια. Η γνώμη των πολιτών δεν υπάρχει, οι πολίτες το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν είναι διαδηλώσεις, δεν υπήρξε καμία επίσημη διαβούλευση μαζί τους. Αν κάποιος έχει αμφιβολίες και το λέω αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έλεγε και ο κύριος Μπαλόνε, θα τους παραπέμψω στη δίκη του Κάφκα, αλλά και στην αλήκη στη χώρα των θαυμάτων. Γιατί συνεχίζουμε εμείς να ασχολούμεθα και να απασχολούμεθα με ακροάσεις, με συζητήσεις κτλ. Εγώ πήγα στο κουμπινόρο, βλέπετε πως έχει η κατάσταση Βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία μεταχείριση, απλά εναπόθεση των απορριμμάτων. Λοιπόν, τα δείχνουμε αυτά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πλήρης παραβίαση όλων των ισχυουσών οδηγιών. Σχετικά με τη Φαλκονιάνα έχουμε εδώ κάποια, κάποιες φωτοτυπίες αυτή ήταν η κατάσταση στη Φαλκανιάνα εδώ και λίγα χρόνια. Υπήρχε μια πάρα πολύ μικρή χωματερή και σιγά σιγά αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε και έγινε αυτό το οποίο βλέπετε. Χωρίς άδειε, χωρίς αδειοδοτήσεις. Και ας μιλήσουμε και φτάνω στο τέλος με την άμα σαλάρια. Πρόκειται για έναν χώρο ο οποίος εντοπίστηκε εδώ και 20 χρόνια και ο οποίος ε, άρχισε να λειτουργεί εδώ και λίγα χρόνια. Για την άμα σαλάρια δεν έχω να σας δείξω κάτι ε, περαιτέρω. Ε, πρόκειται για προβλήματα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων πολιτών και των ηλικιωμένων. Είναι απαράδεκτο ε, να γίνονται αυτά τα ε, προβλήματα, τα μοιάσματα και οι άσχημες μυρωδιές κάνουν ε, μαρτύριο την καθημερινότητα των πολιτών. Ας σταματήσουμε τα κόλπα, ας σταματήσουμε τις ταχυδακτηλουργίες όπως λένε οι Νεαπολιτάνοι. Ας δώσουμε απαντήσεις. Αν υπάρχει Ευρώπη ας κάνει κάτι. Σας παρακαλώ πολύ λέει μη χειροκροτάτε. Ο κύριος Αντωνιώτσι. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να, χαμηλώσετε και αυτές ε, τις... Ε, ε, αυτά τα πανό, καταλαβαίνουμε ποια είναι τα μοιάσματα της ε, περιοχής, τα γνωρίζουμε. Κύριε Αντωνιώτσι, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω γιατί δεχτήκατε να ακολουθήσουμε την διαδικασία του κατεπήγοντος ε, για την περίπτωση της Φαλκονιάνα, θέμα το οποίο βεβαίως εντάσσεται στο γενικότερο σύστημα διαχείρισης ε, απορριμμάτων και που σχετίζεται βεβαίως ε, και με την ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση που επικρατεί στην Ρώμη, στην πρωτεύουσα της Ιταλίας και στην ευρύτερη περιοχή. Η αρχική φωνή έχει γίνει πλέον κραυγή, αλλά δυστυχώς παραμένει αναπάντητη. Γνωρίζουμε, βλέπουμε ε, τους ε, ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, ε, τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ήρθαν εδώ στις Βρυξέλλες έτσι ώστε να μας πούνε τι συμβαίνει εδώ και χρόνια στη χώρα μας και κυρίως στην περιφέρεια της Φαλκονιάνα. Ειλικρινά κυρία Πρόεδρε πρέπει να πω ότι είναι φρικιαστικό που βρισκόμαστε εδώ για μία ακόμα φορά. Για μία ακόμα φορά να προστρέχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για μία ακόμα φορά να προστρέχουμε στην ε, Επιτροπή μας εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αυτά ο πρόεδρος, ε, ο περιφερειάρχης της, ε, του Λάτσιο, ο δήμαρχος της ε, Ρώμης, όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι οι οποίοι με μεγάλη ελαφρότητα και κυρίως εν είδη ποντίου πιλάτου ένυψαν τα σχήρας τους και πέρασαν όλες τις αρμοδιότητες τον ειδικό επίτροπο, ο οποίος επανειλημμένα ε, ε, παίρνει αποφάσεις οι οποίες διαψεύδονται περίτρανα από την συνέχεια των ε, πραγμάτων. Το είδαμε στην περίπτωση του Πιάντε Λόλμο. Είχε πάρει απόφαση σχετική ο Επίτροπος Σωτήλε, αλλά παρόλα αυτά είδαμε ότι στην ουσία ήταν ένας γίγαντας με πύληνα πόδια και βεβαίως κατακριμνίστηκε όλο αυτό το οικοδόμημα δόμημα που είχε δημιουργήσει υποτίθεται ο Επίτροπος Σωτήλε. Ε, αναφερθήκαμε προηγουμένως ε, στην καυκική παράνοια, στη δίκη του Κάφκα, στην αλήκη στη χώρα των θαυμάτων. Όλα αυτά τα λέμε ακριβώς για να δείξουμε την αδυναμία που έχουν ε, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών απέναντι στην κατάσταση αλλά και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σηκώνει τα χέρια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να σταματήσει τη διαδικασία της φαλκο δεν έχουν με κανένα τρόπο γίνει ε, εφαρμοστή ε, ε, οι προβλέψεις και οι διατάξεις των νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε πρόκειται για μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, είτε πρόκειται για μελέτη βιωσιμότητας κτλ. Νομίζω ότι το θέμα είναι Σαφές. Δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα άλλο. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Σας ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε γιατί πραγματικά ε, θελήσατε να αντιμετωπίσουμε εδώ το ζήτημα και γιατί έχετε την ευήκονούση σε όλες ε, τις κινήσεις των ε, πολιτών της Ιταλίας. Δεν θα έπρεπε τα πράγματα να είναι έτσι όμως. Δεν θα έπρεπε για μία ακόμα φορά να προστρέχουν οι πολίτες στη δικιά μας Επιτροπή έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν ζητήματα τα οποία είναι τόσο προσφυλή ε, σε όλους τους ε, πολίτες και τα οποία είναι απαραίτητα έτσι ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να ζήσουν ε, σε ένα υγιές περιβάλλον. Και πραγματικά δεν δέχομαι αυτές τις ασάφειες και τις γενικολογίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατανοήσει ότι έχει όλα τα στοιχεία και όλα τα εργαλεία και όλες τις δυνατότητες στα χέρια της έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει ε, αυτές τις καταστάσεις. Δεν θα θέλαμε για μία ακόμα φορά να, ε, να έρθουμε ε, εδώ σε αυτή την Επιτροπή, για μία ακόμα φορά να καταδικάσουμε καταστάσεις ανεπίτρεπτες στην χώρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφα Αντωνιώτση, λέει η ευχαριστώ πολύ σε όλους τους παρεμβαίνοντες συναδέλφους. Τρέφομαι τώρα σε αυτούς οι οποίοι κατέθεσαν τις αναφορές να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχάς ότι δεν είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι μπορεί να λύσει το θέμα που έχει δημιουργηθεί το θέμα με το Κοινοβούλιο, παραπέμποντας το θέμα πάντα στις εθνικές αρχές. Όταν οι πολίτες στρέφονται σε εμά, το κάνουν αυτό γιατί στα πλαίσια της αρχής της επικουρικότητας, αφού έχουν εξαντλήσει όλα τα επίπεδα αρμοδιοτήτων τοπικών και εθνικών, φτάνουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ζητούν να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάρα πολύ σωστά έχει τη δυνατότητα να παρέμβει όταν οι ε, διαδικασίες λήψης αποφάσεων έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Όπως είπα και στην προηγούμενη αναφορά, δεν έχει νόημα να δίδουμε απαντήσεις αν δεν είναι το επίπεδό μας. Η Επιτροπή γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στο Λάτιο και σε άλλες περιοχές της Ιταλίας. Επανειλημμένα με συναδέλφους αυτής εδώ της Επιτροπής είχαμε την δυνατότητα να ρίξουμε φως στις περιοχές αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν κρίσεις γνωρίζει καλά ποια είναι η κατάσταση, έχει ξεκινήσει πολλές διαδικασίες επί παραλήψη, επί παραβάση, έχουν επίσης οδηγηθεί την Ιταλία και στο δικαστήριο για τα θέματα αυτά. Στην έκθεση που είχαμε διατυπώσει στα πλαίσια της τελευταίας επίσκεψής μας εκεί, υπό την καθοδήγηση της κυρίας Μέρκης, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συγκεκριμένες ε, δράσεις. Εδώ και ένα χρόνο το κάναμε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα λέει ότι τελικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν ολοκληρωθεί η Ιταλική Εθνική Διαδικασία. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να παραμείνουμε πάντα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ζητάμε μία παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία να μην είναι μόνον και αποκλειστικά μία παρέμβαση επιβολής κυρώσεων. Το να επιβάλλει κανείς επιπλέον κυρώσεις δεν χρησιμεύει σε τίποτα από το άλλο από το να χειροτερεύει η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Πρέπει να γίνουν σεβαστά τα περιεχόμενα της οδηγίας. Πρέπει να υπάρξει παρέμβαση ακόμα και σε προληπτικό επίπεδο, χωρίς να αποκλείσουμε κάποιες μορφές ε, λύσης. Εγώ λοιπόν ζητώ από τους συναδέλφους ε, ε, να συμφωνήσουν ότι θα πρέπει να παραμείνουν φυσικά ανοιχτές αυτές οι αναφορές και θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα με μεγαλύτερη ευαισθησία. Μεταφέρω προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία πρόσκληση η οποία έχει γίνει επανειλημμένα στο παρελθόν ε, και από τις συναδέλφους Άουγκεν και Μέρκης. Αποστέλουμε λοιπόν μία πρόσκληση προς τον Επίτροπο Ποτότσνικ να πάει στην Ιταλία, να δει πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας, αλλά να προσπαθήσουμε να παρέμβουμε με μια αναπλήρωση, αν θέλετε, ε, της ε, ε, εκτελεστικής διαδικασίας. Ξέρετε ότι εμείς έχουμε ένα ειδικό επίτροπο στην Ιταλία που ασχολείται με το θέμα όταν είναι ε, έτσι η κατάσταση, όταν δηλαδή υπάρχει διορισμός ειδικού επιτρόπου, καλύτερα να το αναλαμβάνει ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, παραμένουν ανοιχτές οι αρμοδιότητες αυτές. Θέλει ένα λεπτό επιπλέον η κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε η παραδοσιακή θα έλεγα συμπεριφορά ε, ε, ενός από τους αναφέροντες ο οποίος ε, κυκλοφόρησε με ένα κάτι το οποίο δημιούργησε ένα άσχημο, μια άσχημη μυρωδιά. Αυτή η άσχημη μυρωδιά δεν έχει τίποτα με αυτό που μυρίζουν οι άνθρωποι στο Κουπινόρο, στη Φαλκονιάνα και κυρίως στην Άμα Σαλάρια οι άνθρωποι στους χώρους κατοικίες τους, οι άνθρωποι στους χώρους εργασίας τους βλάπτονται συστηματικά από τέτοιου είδους παρενοχλήσεις. Λοιπόν, ήταν δύσκολο αυτό που συνέβη, αλλά παρόλα αυτά οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν φωνή, μόνο υπογραφές μαζεύουν και μόνο διαμαρτύρονται. Πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσουμε την πρόεδρο Ματσόνη για την ευαισθησία την οποία επέδειξε και ε, πράγματι θεωρούμε ότι είναι πρωταγωνίστριά μας στον τομέα αυτό, η σημεοφόρος μας. Ευχαριστώ κύριε Αντζελίλη. Λοιπόν, παραμένουν ανοιχτές οι συγκεκριμένες ε, αναφορές, αλλά σημειώνω εκ νέου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την ανάγκη για μια διαφορετικού τύπου και πνεύματος μορφή συνεργασίας με το Κοινοβούλιο και τους αναφέροντες. Οι συνάδελφοι όλοι συμμερίζονται αυτό το οποίο λέγω. Πρέπει η Επιτροπή να πάει στην Ιταλία, να έρθει μαζί μας στην Ιταλία και να προσπαθήσει να παρεμβαίνει πλην το πρόβλημα καταστεί πλήρως άλυτο. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και την κυρία Αντζελίλη που ζήτησε συγγνώμη για συμπεριφορές που απάδουν της παράδοσης του Ιδρύματός μας και τελειώνουμε κλείνοντας την αναφορά 18. Μη χειροκροτείτε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εγκαταλείψετε την ε, αίθουσα χωρίς φασαρία, ε, γιατί έχουμε ήδη αργοπορήσει. Φτάνουμε στο επόμενο σημείο. Είναι η αναφορά 51 2013 του κυρίου Πέντρο Χιμένεθ Σαν Χωσέ, Ισπανικής Ιθαγένειας, που απευθύνεται στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να καταγγείλει ε, κάποιες παρανομίες όσον αφορά δραστηριότητες εξόριξης, αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή Ντονιάνα Ουέλβα, περιοχή που προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000. Για την αναφορά αυτή θα δώσω τον λόγο στον υπογράφοντα μάλλον τον εκπροσωπούντα τον, ε, ε, ε, τον αναφέροντα, τον κύριο Σμιθ Χάμερστάιν. Is Mr. No. Sorry. The floor. Can you help me? Mr. Jimenez. Mr. Jimenez señora presidenta. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να γίνει λίγη ησυχία. Εν πάση περιπτώσει, πριν μπω στα πιο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την αναφορά, να σας παρουσιάσω το πλαίσιο, θα έλεγα. Αναφερόμεθα σε μια περιοχή, στην περιοχή της επαρχίας της Κουέλβα και σε έναν προστατευόμενο χώρο, το πάρκο ακριβώς της Ντονιάνα. Στην περιοχή ε, του Καντίζ, της Κουέλβα και της Σεβίλη. Η περιοχή της Χουέλβα ήδη από τη δεκαετία του 60 και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φρανκό είχε έναν βιομηχανικό πόλο, χημικό, που παρήγαγε πάρα πολλά προϊόντα τα οποία μόλυναν το περιβάλλον και η Χουέλβα αντιμετώπισε ε, μόνιμα επεισόδια ε, προβληματικά για το περιβάλλον η προστασία του περιβάλλοντος εκείνη την εποχή ήταν ανύπαρκτη, εν πάση περιπτώσει πολύ ελευθεριακή αν θέλετε, δημιουργήθηκαν προβλήματα μόλυνσης των υδάτων και στα ποτάμια και ε, στη θάλασσα υπήρξε επιμόλυνση των ε, ε, υδάτινων πόρων της περιοχής Υπήρξε επίσης ε, μια, ε, μια, ένα μέρος εναπόθεσης ε, χημικών φωσφορούχων, πρόκειται για το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Ευτυχώς και χάρη και στις δικές σας εργασίες τελικά σταμάτησε η τροφοδοσία αυτού του, του τόπου της χωματερής για τα χημικά αν θέλετε ε, έχουν εναποτεθεί 120 εκατομμύρια τόνοι φωσφορούχων, λέει ο μιλητής εκεί. Por tanto, de una Μιλάμε για μια περιοχή όπου τα τελευταία χρόνια πέρα από τον βιομηχανικό αυτό πόλο, χημικό βιομηχανικό που ε, κατασκευάστηκε ε, το 1960 δημιουργήθηκε και ένας πόλος ενεργειακής παραγωγής, ένα εργοστάσιο παραγωγής θερμικής, ε, ε, μέσω, ένα θερμικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 35 ΜΒ, 2 χιλιόμετρα επίσης ένα νέο τέτοιο εργοστάσιο από το παλαιό διευρύνθηκε η εναπόθεση φυσικού αερίου και η εκμετάλλευση φυσικού αερίου, δημιουργήθηκε ίσως η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής βιομάζας, φυσικού αερίου από βιομάζα. Ε, γενικά υπάρχει συμπαραγωγή λοιπόν από όλες αυτές τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Υπάρχει επίσης και ένα δηληστήριο που πέρασε από 5 εκατομμύρια πετρέλαιο τόνους έχει φτάσει τώρα στα 9. Λοιπόν αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι έχουμε να, να κάνουμε με μια περιοχή η οποία απειλείται από το περιβάλλον της ήδη από την εποχή της δικτατορίας του Φράνκο και ακριβώς δεν έχουν γίνει προσπάθειες ε, ε, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λόγω ακριβώς της υπερσυγκέντρωσης αυτών των χημικών βιομηχανιών και η κατάσταση έχει πλέον χειροτερεύσει. Ε, και μάλιστα πρόκειται για τη μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή της Ισπανίας, το πάρκο της Ντονιάνα, μιλάμε για ένα καταφύγιο ίσως και το μεγαλύτερο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο της ε, Ισπανίας. Πρόκειται για μια ε, είναι σαφές ότι στην Ανδαλουσία υπάρχουν όλων των ειδών τα προστατευόμενα συστήματα, όχι μόνο μέσω των οδηγιών των ευρωπαϊκών, των εθνικών, αλλά μέσω και των περιφερειακών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα προστασίας του πάρκου της Ντονιάνα, και της κοινοτικής οδηγίας την οποία παραπέμπουμε εμεί στα πλαίσια της αναφοράς μας και δεν είναι απαραίτητο στα πλαίσια αυτής της σύντομης παρουσίασης να αναφέρω. Εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι να πούμε ότι πρόκειται για μια ζώνη η οποία υπόκειται σε όλες τις μορφές προστασίας που υπάρχουν στα πλαίσια της περιφερειακής διοίκησης. Ένα καταφύγιο λοιπόν της φυσικής ζωής που πρέπει να προστατεύσουμε και έχει γίνει αντικείμενο προσοχής και των ευρωπαϊκών οργάνων και έχουν υπάρξει επενδύσεις για την προστασία της φύσης, έχουν γίνει επενδύσεις για την αποκατάσταση των ζημιών λόγω των δραστηριοτήτων στα πλαίσια της αηφορίας και παρόλα αυτά συζητάμε όπως λέμε στην αναφορά μας για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει μόνο σαν στόχο την παραγωγή φυσικού αερίου αλλά κυρίως την αποθήκευση αυτού του φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ζώνη η οποία είναι στην περιοχή αυτή όπου εξάγεται το φυσικό αέριο και την δημιουργία ε, ενός αγωγού αερίου 18 χιλιόμετρων ε, που θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα, ένα πολύ μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο. Μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο είναι απαράδεκτο, ένα σχέδιο που παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ισπανική νομοθεσία. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτραπεί να προχωρήσει ένα τόσο απαράδεκτο σχέδιο όπως αυτό. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και το Συμβούλιο στην Τονιάνα το οποίο εξεφράστη θετικά προεδρεύεται από τον Φελίπε Γκονσάλες, τον τέος πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος ε, παρουσιάζοντας ε, την παρέτηση του Συμβουλίου αυτού συμμετέχει ακριβώς στο Διοικητικό Συμβούλιο και της επιχείρησης η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ε, εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πάρει όλα τα απαιτούμενα μέτρα έτσι ώστε να γίνει σεβαστή η οδηγία σε περιβαλλοντικό επίπεδο και να αποφευχθεί ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα απαράδεκτο αυθεντικό σκάνδαλο και παρουσιάζει κινδύνους για τους κατοίκους της περιοχής. Εξ ονόματος λοιπόν της Ένωσης Μέσο Ντελαρία Ντεγουέλβα που είναι μια δεύτερη αναφορά αλλά έχει δυστυχώς εκλάθους τον ίδιο αριθμό με την προηγούμενη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Χάμερστάιν. Παρακαλώ να σεβαστείτε τον χρόνο γιατί δεν έχουμε ε, δυνατότητα μεγάλη χρονικά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκπροσωπώ την Μέσα Ντελαρία που είναι μια ένωση πολιτών, όχι μια πολιτική οργάνωση η οποία φροντίζει το περιβάλλον στην περιοχή της Βουέλβα. Πράγματι μιλάμε για δύο αναφορές διαφορετικές η μία από την άλλη. Από τη μία υπάρχει μία αναφορά στην οποία αναφέρθηκε ο Προλαλήσας που αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο ε, πρόγραμμα και πράγματι ε, ένας από τους πολιτικούς εκπροσώπους που είναι εδώ συμμετέχει στην περιφερειακή κυβέρνηση που είναι υπεύθυνη για να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις. Αυτό είναι ε, θα έλεγα κάτι το οποίο ε, εκπλήσει, είναι ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να ειδωθεί. Τώρα σχετικά με την δική μου αναφορά της Μέσα Λαρία αφορά την εξαγωγή φυσικού αερίου της Ρεψόλ, όχι φυσικού αερίου, ε, που δραστηριοποιείται στην περιοχή αυτή ε, εδώ και αρκετά χρόνια χωρίς σεβασμό των τοπικών ε, ισχυουσών ρυθμίσεων και την εναπόθεση φωσφορούχων σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση χωρίς να σέβεται αυτά τα οποία έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δική σας Επιτροπή ότι θα πρέπει δηλαδή η επιχείρηση αυτή να παρουσιάσει ένα σχέδιο καθαρισμού της περιοχής από τις εναποθέσεις φωσφορούχων. Έχουμε να κάνουμε στην περιοχή με λίγα λόγια με ένα Wild West, με την άγρια δύση την περιβαλλοντική. Λειτουργεί επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη επίσημη άδεια. Η τοπική κυβέρνηση λοιπόν συνεχίζει να δέχεται να γίνονται ζημιές οικολογικές στην Χουέλβα και στο Περιφερειακό Πάρκο της Ντονιάνα. Όπως και να έχουν λοιπόν τα πράγματα, στην περίπτωση ε, της ε, υπόθεσης του φυσικού αερίου περιμένουμε ε, κάποιες απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση της Ρεψόλ και με τη μόλυνση που έχει δημιουργήσει η εταιρεία αυτή, η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας γνωρίζει ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη βιομηχανική δραστηριότητα που δεν είναι συμβατή με την κοινωνική νομοθεσία, που δεν έχει αδειοδοτηθεί από κανέναν. Σύμφωνα, δεν σέβεται την οδηγία λοιπόν για, την, τον καθαρισμό των εδαφών εκμετάλλευσης και αυτή τη στιγμή η επιχείρηση αυτή λειτουργεί, συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς άδεια και έχει δημιουργήσει τεράστιες εναποθέσεις ε, ουσιών που μολύνουν και τα ύδατα της περιοχής γύρω από την Χουέλβα και δεν λειτουργεί με βάση την ενιαία περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τον τοπικό και κοινοτικό νόμο. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα δημιουργηθεί στο μέλλον, μιλάμε για ένα υπάρχον θέμα, μιλάμε για μια δραστηριότητα με εκατοντάδες εργαζομένους, με χιλιάδες φορτηγά από τη δεκαετία του 90, χωρίς, είπαμε, αδειοδότηση, χωρίς ε, μελέτες και κτλ. Είναι μια κατάσταση λοιπόν πάρα πολύ απογοητευτική, ανησυχητική. η Ρεψόλ εκμεταλλεύεται την ε, εξαγωγή φυσικού αερίου με βάση παλαιές άδειες του 2004 και 2005 που δεν έχουν ανανεωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και δεν δίνουν δυνατότητες τέτοιες στην επιχείρηση. Δεν έχουμε λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις από την κυβέρνηση την τοπική και αυτό το οποίο ε, μας απασχολεί είναι το συγκεκριμένο σχέδιο λοιπόν της Επιτροπής Ρεψόλ δεν είναι κάτι το οποίο είναι σχετικό με το πρόγραμμα Κάστορ, σαν παράδειγμα της περιοχής του, της ε, περιοχής ε, του Εύρω. Ε, εκεί έχουν λειτουργήσει κάποιες δραστηριότητες με βάση την αδειοδότηση, αλλά στην περίπτωση του προγράμματος Ποζεϊντών η Ρεψόλ λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια εκτός νομιμότητας, χωρίς αδειοδότηση χωρίς την ενιαία περιβαλλοντική αδειοδότηση η οποία απαιτείται ε, για τον καθαρισμό της περιοχής. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές, δηλαδή την περιφέρεια της, την περιοχή της Ανδαλουσίας και την τοπική κυβέρνηση, να φέρουν εις πέρα στις αρμοδιότητές τους, στις υποχρεώσεις τους και για την εξαγωγή αερίου και για την εναπόθεση φωσφορούχων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα σημειώσαμε αυτά. Δεν μπορούμε επί της ουσίας να πούμε πολλά πράγματα γιατί η αναφορά είναι ακόμη σχετικά πρόσφατη, δηλαδή μόλις τον Νοέμβριο την λάβαμε. Την παρακολουθήσαμε, άκουσα προσεκτικά τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι αναφερόμενοι γνωρίζουμε τα προβλήματα της ε, περιφέρειας. Έχουμε και μια διαδικασία προσφυγής ήδη για, ε, για την απόρριψη ε, φωσφορούχων και οι δύο αναφορές είναι συνδεδεμένες. Όσον αφορά το πρόβλημα του φυσικού αερίου θα εξετάσουμε προσεκτικά την αναφορά και θα απαντήσουμε στο, σε έφθετο χρόνο στην Επιτροπή Αναφορών. Κύριε Τουργκάης, εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή έχουμε και τις δύο αναφορές, να κάνουμε το ίδιο όπως κάνουμε κάθε φορά όταν έχουμε και τους αναφερομένους, όπως ε, όταν έχουμε και τις δύο πλευρές. Έχουμε και τους αναφερομένους από την, έχουμε και την πλευρά των επιχειρήσεων μάλλον. Κύριε Πρόεδρε, να ακούσουμε δηλαδή και αυτούς, ώστε να ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Sí, una, una de las dos empresas, sí. Μάλιστα, μία από τις δύο επιχειρήσεις φαίνεται πως είναι παρούσα. Λοιπόν, λέει η Πρόεδρος, είχε ανακοινωθεί η παρουσία εκπροσώπων της ε, εταιρείας έχει συμβεί και στο παρελθόν να δώσουμε και στο άλλο μέρος τον λόγο. Πάντως θα ήθελα να... Επομένως, ναι, μπορούμε να δώσουμε τον λόγο, αλλά πραγματικά επειδή έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, θα ήθελα να σας ζητήσω μέσα σε δύο λεπτά να αναφερθείτε στη δικιά σας τοποθέτηση. one moment. Ah, Ένα λεπτάκι για λόγους μεθοδολογίας. Νομίζω ότι μέχρι τώρα οποτεδήποτε στην Επιτροπή μας έχουμε ε, αναφορά, είχαμε μόνο τους ε, αναφερόμενους. Μονάχα όταν ε, είχαμε περιπτώσεις όπου εμπλέκοντο δημόσιες υπηρεσίες, δίναμε το λόγο στο άλλο μέρος που ήταν η δημόσια υπηρεσία. Εδώ έχουμε ιδιωτική ε, ε, ε, ιδιωτική εταιρεία βεβαίως καταλαβαίνουμε είμαστε όλοι πολιτισμένοι άνθρωποι μπορούμε να το κάνουμε να δώσουμε το λόγο για λίγο αλλά δεν έχει γίνει μέχρι τώρα Πρόεδρος, ναι, ε, ίσως έχει δίκιο ο συναδελφός Μεγέρα, αλλά νομίζω ότι το έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, ε, ήδη είχα ζητήσει και εγώ από τους καλεσμένους μας ε, να είναι πάρα πολύ σύντομοι έτσι ώστε να, δώσουν τον, ε, να δώσουμε τον λόγο ξανά και στους αναφερόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Πάκο Βελάσκο και εργάζομαι στην εταιρεία φυσικού αερίου Μπένοσέρ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Λοιπόν, ήδη βλέπετε εδώ μια πρώτη διαφάνεια όπου περιγράφεται το σχέδιο. Στην ουσία θέλουμε να αντικαταστήσουμε ε, κάποιες από τις υφιστάμενες ε, υποδομές ε, έτσι ώστε να προωθήσουμε την παραγωγή φυσικού αερίου μέσα από νέους αγωγούς. Επίσης προβλέπουμε και την υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου. Εδώ και 30 χρόνια βεβαίως βρισκόμαστε στην περιοχή και ασχολούμαστε με την ε, εξόριξη αερίου. Κατά την άποψή μας ε, δεν υπάρχει καμία παραβίαση του, του, της ενωσιακής νομοθεσίας. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να σας πω ότι η Οδηγία 92, ε, καθώς επίσης και η Οδηγία για την προστασία των πτηνών, γίνονται απολύτως σεβαστές. Επίσης δεν υπάρχει καμία παραβίαση της Ράμσα το φυσικό αέριο εκεί συναντάται με φυσικό τρόπο. Ε, θεωρούμε επίσης ότι το πρόγραμμα αυτό δεν είναι ασύμβατο με το δίκτυο Natura 2000. Δεν θίγεται ε, το εσωτερικό του Εθνικού Πάρκου, αλλά μόνο οι περιβάλλοντες φυσικοί χώροι έχει υπάρξει μια εξαντλητική ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 7 χρόνια. Έχουμε κάνει πάρα πολλές μελέτες, είμαστε νομίζω συμβατοί με την οδηγία. Έχει υπάρξει επίσης και δημόσια διαβούλευση. Έχουν εφαρμοστεί πάρα πολλά μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στην δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχουν υπάρξει εργασίες επίσης ε, για την αποκατάσταση του χώρου και την προστασία της πανίδας και της ε, χλωρίδας. Όλα αυτά είναι εκτός ε, του πάρκου και στην ουσία είναι κάτι το οποίο καλύπτει τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Είναι συμβατό επίσης και με τα χωροτεκτικά σχέδια της περιοχής αυτής και την προστασία των φυσικών περιοχών και της προστασίας του πάρκου της Ντονιάνα. Όπως έχουν πει οι υπεύθυνε αρχές για τα θέματα αυτά. Τέλος, δεν πρόκειται για μια βιομηχανική δραστηριότητα ή για την αύξηση μιας βιομηχανικής δραστηριότητας. Δεν είναι μια δραστηριότητα. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Βλέπετε τον υπάρχοντα, την υπάρχοντα, υπάρχουσα ρύθμιση. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι αν δεν προχωρήσει ε, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό θα είναι αρνητικό και για την περιοχή και για την χώρα. Θα δημιουργηθεί επίσης και ζημία φυσικά στην ε, επιχείρησή μας. Μπορείτε να καταθέσετε αν θέλετε και την τεκμηρίωση την οποία έχετε φέρει. Θα είναι καλό και για την ε, εργασία μας. Ένα λεπτό ε, στον καθένα, στους ε, αναφέροντες. Δίνω πρώτα το λόγο στον ε, κύριο Χιμένες. Δεν θέλει Για μια στιγμή. Έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Μέγερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου φαίνεται ότι η συγκεκριμένη αυτή αναφορά λόγω ακριβώς του χώρου στον οποίο αναφερόμεθα, μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος γίνεται αντικείμενο προστασίας και εφαρμόζονται οι αρχές επίσης ε, της πρόληψης που πρέπει να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο στις ευρωπαϊκές οδηγίες, στο δίκτυο Natura 2000 και στα επιμέρους ε, τοπικά προγράμματα αλλά και αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση του προγράμματος Κάστορ. Ε, αυτή η εκμετάλλευση προκάλεσε σεισμικές συνέπειες και όταν κυκλοφόρησε από πλευράς του Υπουργείου η μελέτη ε, ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων χωρίς κινδύνους υποτίθεται ε, βλέπουμε ότι προβλέπεται τελικά η δυνατότητα σεισμικής αντίδρασης. Άκουσες φυσικά, άκουσα τους εκπροσώπους της ε, ιδιωτικής εταιρείας, κατάλαβα ότι αυτές, ε, αυτά τα οποία είπε είναι εξαιρετικά. Μιλάμε όμως για κάτι τελικά το πάρα πολύ σοβαρό στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι αλήθεια ότι εμείς οφείλουμε, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλωστε, να ασχοληθούμε στο μέλλον με την συγκεκριμένη αυτή πρόσφατη αναφορά. Εγώ έχω θέσει ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά και θα πρέπει επίσης να μεταφερθεί ε, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος η ανησυχία μας έτσι ώστε να συμπεριληφθεί μια μελέτη για τις πιθανές σεισμικές αντιδράσεις αυτού του είδους στην δραστηριότητα και σε σχέση με το πρόγραμμα Καστόρ το οποίο ακύρωσε ουσιαστικά ένα μεγάλο τμήμα του προγράμματος και απαιτείται, είναι προαπαιτούμενο, εν περιπτώσει, να υπάρξει ε, μια τέτοια ε, σεισμική μελέτη. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά, έτσι θα συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες και εμείς απλά να στείλουμε μια επιστολή, να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας και να απαιτήσουμε στο εσωτερικό της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να υπάρξει και μελέτη σεισμολογική. Ο κύριο Ιτουργκάης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ζητήσει πληροφορίες από τις Ισπανικές Αρχές και τις έχει πάρει. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ισπανίας έχει δώσει συμπληρωματικά στοιχεία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να σημειώσω τρία στοιχεία από, αυτές τις, από αυτή την τεκμηρίωση. Πρώτον, οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης των προγραμμάτων βασίζονται στον αναφερειμένο νόμο του 2011. Και επίσης είναι συμβατό το πρόγραμμα και με το δίκτυο Natura 2020. Έχει υπάρξει ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό πλαίσιο για την εφαρμογή του προγράμματος. Και τρίτον, οι μελέτες ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων ε, αναφέρονται σε συγκεκριμένα προγράμματα δηλαδή οι τοπικές ε, ε, αρχές όπως επίσης και οι τοπικές κυβερνητικές αρχές εκφράστηκαν με ε, ολοκληρωμένα προγράμματα για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες καταλήγοντας το ότι δεν θα υπάρξουν ουσιαστικά προβλήματα για το Natura 2020. Συνεπώς λοιπόν όχι μόνο η κεντρική κυβέρνηση αλλά και η κυβέρνηση η περιφερειακή της Ανδαλουσίας κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα με αυτά στα οποία κατέληξε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα πρέπει λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των πιλωτικών προγραμμάτων και υπό το φως των συμπληρωματικών πληροφοριών να μας κρατήσει ενήμερους. Ευχαριστώ κύριος Γιάννης. Εγώ χαίρομαι που λειτουργεί ε, προληπτικά η γραμματεία και η πρόεδρος της Επιτροπής. Εγώ δεν ζήτησα το λόγο, αλλά ξέρετε ε, να αναγνωρίζετε αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το θέμα και για τα συμφέροντα της περιοχής τους, της Εβίλης δηλαδή και της επαρχίας αυτής. Δεν είχα ζητήσει το λόγο για έναν πάρα πολύ απλό λόγο και πολύ γνωστό θα έλεγα. Εγώ ήρθα εδώ να ακούσω, δεν ήρθα να πω κάτι, δεν έχω κάτι να πω. Θα άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά αυτά που είπαν και οι αναφέροντες και η Επιτροπή και η επιχείρηση και θα τα λάβω υπόψη μου. Ενημερώθηκα πρόσφατα για τη συγκεκριμένη αναφορά σχετικά με τη θέση της κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Όχι μόνο γιατί το δικό μου κόμμα και το κόμμα του Βίλη συμμετέχουν στην κυβέρνηση, αλλά είναι θα έλεγα το επίπεδο εξουσίας το πιο κατάλληλο για να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Μιλάμε βέβαια για μια περιοχή η οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη περιβαλλοντικά και θα πρέπει να δώσουμε τις απαιτούμενες εγγυήσει και διασφαλίσεις έτσι ώστε να μην φυγεί το περιβάλλον στην περιοχή. Ευχαριστώ κύριε Γιάννης. Ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς να βάλω σε ένα πλαίσιο το τι είναι πραγματικά η Ντονιάνα, να ενημερώσω ότι πρόκειται πράγματι για μια περιοχή η οποία εκπλήσει με τον φυσικό της πλούτο και τη φυσική της ποικιλία. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες ανάπτυξης στην περιοχή αυτή και σε επίπεδο οικιστικό και σε επίπεδο κτηριακό και σε επίπεδο βιομηχανικό. Όπως είπαν ε, ο εκπρόσωπος της περιοχής, αυτό μπορεί να είναι κάτι το θετικό όχι μόνο για την περιφέρεια αλλά και για το σύνολο της χώρας. Έχουμε να κάνουμε με ένα σημαντικό οικονομικό περιπτώσει διακύβευμα ε, και σε επίπεδο όμως σημαντικό είναι και το περιβαλλοντικό αντίστοιχο. Από αυτά που άκουσα από τους αναφέροντες έχω την αίσθηση ότι στην Τονιάνα και στην Ανδαλουσία τα θέματα του περιβάλλοντος δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Αν και βέβαια ε, υπάρχουν κάποιες, εγκαταστά, κάποιες εγκαταστάσεις βιομηχανικές, υπάρχουν επενδύσεις στον τομέα αυτό σχετικά με το προηγούμενο θέμα το οποίο ε, συζητήσαμε για την Ιταλία βλέπουμε ότι τα πράγματα μπορεί να μοιάζουν λίγο και στην ε, δική μου χώρα. Αυτά τα οποία μας είπαν ε, οι Ιταλοί αναφέροντες είναι θα έλεγα ένα θέμα το οποίο αφορά και τον νότο της Ισπανίας. Είδαμε ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει και ένα θέμα με τη συμμετοχή στη λήψη των διαδικασιών του Φελίπε Γκονσάλες. Πρέπει να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες και σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσει και από την Ισπανική κυβέρνηση και από τις περιφερειακές κυβερνήσεις οι οποίες υποτίθεται πρέπει να είναι πρωταγωνιστικές για το σεβασμό του περιβάλλοντος να έχουν πάντα ένα συγκεκριμένο στόχο ε, να προωθήσουν τα τοπικά συμφέροντα, τα συμφέροντα των πολιτών και τα συμφέροντα της προστασίας του περιβάλλοντος γενικά. Ε, thank you and... Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη για την ε, έλλειψη προσοχής στιγμιαία ε, ήρθε η κυρία Ορέιλι, η Ευρωπαία Διαμεσολήτρια, η οποία θα πάρει το λόγο αργότερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό και επομένως θα δώσω τώρα το λόγο για ένα λεπτό στον Πέδρο Χιμένε Σαγκοσέ για την απάντηση. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι πολιτικός εκπρόσωπος δεν είμαι πολιτικός εκπρόσωπος, εκπροσωπώ βέβαια καμία επιχείρηση ή κανένα πολιτικό χώρο συγκεκριμένο, αλλά τους πολίτες. Και ήθελα να προσπίσω μια άποψη η οποία είναι ταυτόσιμη με αυτή που έχουν όλες οι οικολογικές οργανώσεις στην Ιταλία σε σχέση με το περιβάλλον. Εγώ άκουσα αυτά τα οποία είπε η επιχείρηση, η οποία προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα, και είπε ότι ακριβώς ένας από τους στόχους είναι η μεγιστοποίηση των κερδών και λέγει ότι η αδειοδότηση του συστήματος αυτού που λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια θα πρέπει να ελέγχεται βέβαια και περιβαλλοντικά, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και γι' αυτό η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Αυτό το οποίο υποστηρίζει η επιχείρηση είναι να αυξήσει ακριβώς τον αριθμό των, ε, των σημείων στα οποία εν θα γίνεται η εξόριξη και να οικοδομήσει ένα νέο αγωγό φυσικού αερίου άνω των 18 και χιλιόμετρων και θέλει ακριβώς να διατηρήσει και τα, τους χώρους ε, που έχει προχωρήσει στην ε, εξαγωγή του φυσικού αερίου για αποθήκευση ποσοτήτων. Ε, θα πρέπει ακριβώς για να προχωρήσουμε να υπάρξουν μελέτες που θα επιτρέψουν την αποθήκευση και του διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών η οποία έχει παίξει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος και για την εναπόθεση των φωσφορούχων και να εκφράσω την ανησυχία μου για κάποιες πολιτικές προτάσεις οι οποίες τίνουν στην εξασθένιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής της Επιτροπής σας. Για το θέμα το οποίο μας απασχολεί σήμερα θα ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα Ποσειδών έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια όπως αυτή προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία. Και απαιτώ λοιπόν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυβέρνηση της Ανδαλουσίας να σεβαστούν τις νομικές ρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Παραμένει ανοιχτή λοιπόν η αναφορά όπως το ζήτησαν και άλλοι συνάδελφοι και μετά από αυτά που είπε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιμένοντας δηλαδή περισσότερη ενημέρωση από πλευράς της, εκφράζω την ευαρέσκειά μου για το πνεύμα συνεργασίας το οποίο θα πρέπει να ισχύει ανάμεσα στην Επιτροπή ε, και την δική μας. Κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ τους υπογράφοντες οι οποίοι υπέβαλαν ε, το συγκεκριμένο αυτό σοβαρό θέμα και βεβαίως εμείς είμαστε πάντα εδώ έτσι ώστε να συζητούμε περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία δυστυχώς αντιμετωπίζουμε σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνω το σημείο αυτό και τώρα ε, θα ε, δώσουμε την θέση που τους αρμόζει στους καλεσμένους μας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον πρόεδρο της Ιρλανδικής Επιτροπής Αναφορών στον κύριο Μάκλομ Λάιμ. You can repeat your name in the right way. Thank you. Λυπάμαι, δεν προφέραμε το, το όνομά σας ε, σωστά. Σας καλωσορίζουμε πάντως, εσάς και όλη την αντιπροσωπή. Ε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να εμφανιστούμε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής σας καθώς και για την υποδοχή που μας επιφυλάξατε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την αντιπροσωπεία μου. Με συνοδεύουν τρία μέλη της Επιτροπής. Μάικλ Πίκετ που είναι και αντιπρόεδρος της ε, Ιρλανδικής Βουλής, ο βουλευτής Ήλι Ρέι και η γερουσιάστρια Σούζαν Νοκίφτ. Μας συνοδεύουν επίσης αξιωματούχοι της ε, διοικήσεως της Βουλής. Η Επιτροπή Αναφορών σας είναι υπόδειγμα για το πώς πρέπει να λειτουργεί μια Επιτροπή Αναφορών και στόχος μας είναι να διδαχθούμε από εσά και από τις διαδικασίες που εφαρμόζετε. Ευχαριστώ την γραμματεία σας, ιδίως τον David Lowe που ήρθε στο Δουβλίνο για να μας συμβουλεύσει στην φάση αφετηρίας. Συμβουλές πραγματικά σπουδαίες για την έναρξη του έργου της Επιτροπής μας. Έχουμε αρχίσει από πέρσι το Σεπτέμβριο να εργαζόμαστε στη βάση μιας απλής διαδικασίας όπου ε, άτομο ή ένωση προσώπων μπορούν να απευθυνθούν στην Επιτροπή Αναφορών και των δύο σωμάτων, κοινοβουλευτικών σωμάτων της Ιρλανδίας. με σεβασμό των συνήθων κοινοβουλευτικών κανόνων. Βέβαια, η αναφορά δεν ε, μπορεί να αναφέρεται σε υπόθεση πεκρεμωδική. Κατά την εξέταση της αναφοράς ενδέχεται να προσκαλέσουμε τον αναφερόμενο να προσέλθει ενώπιον ημών να λάβει το λόγο Αναζητούμε επίσης γραπτά ή προφορικά στοιχεία από την κυβέρνηση ή από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Μπορούμε επίσης να παραπέμψουμε την αναφορά σε άλλη επιτροπή για να την εξετάσει και να επανέλθει ή να την διαβιβάσουμε στον διαμεσολαβητή ή σε άλλο ειδικό όργανο που έχει ως στόχο να ασχολείται με αυτά. Επίσης την διαβιβάζουμε στους υπουργούς και σε άλλα αρμόδια πρόσωπα. Μετά από την εξέταση των γραπτών και προφορικών στοιχείων που έχουμε λάβει, η Επιτροπή μας, ε, η Επιτροπή αναλαμβάνει απόφαση σχετικά με την δράση που πρέπει να αναλάβει και αναλόγως με τον κανονισμό της Βουλής και της Γερουσίας. Ολοκληρώνω την σύντομη παρέμβασή μου με την επιθυμία να εξηγήσω τη σχέση που έχουμε με το έργο της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, που είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την Έμιλι Ωραίλη, που αποδείχθηκε να είναι από τις σημαντικότερες συμμάχους μας για τα, για την, στον αγώνα υπέρ των δικαίων των πολιτών. Διαθέτει μεγάλη γνώση και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο, στα νέα της καθήκοντα. Θέλαμε να κάνουμε αυτή την πρώτη σύντομη παρέμβαση πριν η κυρία Ορέιλη μπορέσει να σας απευθύνει το λόγο για να σας αναπτύξει τα πεπραγμένα της ως τώρα. Η πρόεδρος Ματσόνη, σας ευχαριστώ πολύ που έχετε έλθει εδώ και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υποστηρίζουμε την κυρία Ορέιλη πάση δυνάμει και είμαστε αποφασισμένες να συνεργαστούμε με την Ευρωπαία Ombudsman, Ombudswoman, αν μπορεί κανείς να το πει έτσι. Ήδη εδώ και μερικά χρόνια αρχίσαμε και σωστά μάλιστα και να συνεργαζόμαστε με τον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή και είμαι βεβαίω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο έτσι ώστε η συνεργασία μας να είναι ενδιαφέρουσα. Αρχίζουμε με την ειδική έκθεση που θα παρουσιάσει τώρα η κυρία Ορέιλι και που έχει ιδιαίτερη ευαισθησία. Και πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή της συνεργασίας μας. Καλή αρχή. Και πραγματικά προμηνύεται καλά, καλούς ιονούς για την εργασία της κυρίας Ορέιλη. Ευχαριστώ και πάλι. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Ορέιλη. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει η κυρία Ορέιλη, αξιότιμες κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι η πρώτη μου ευκαιρία που απευθύνω το λόγο στους Ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πρώτα τους Ευρωβουλευτές που με έδωσαν προηγούμενα φέτος την σημαντική αυτή θέση. Κατανοώ τη σημασία της Επιτροπής Αναφορών για τους Ευρωπαίους πολίτες και ασφαλώς επιθυμώ να ενισχύσω τη συνεργασία μεταξύ του γραφείου μου και της Επιτροπής σας. Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι είμαι ακόμη σήμερα που βρίσκονται σήμερα ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ιρλανδικής Επιτροπής Αναφορών. Παρόλο λοιπόν την χαρά μου που μπορώ να σας απευθύνω το λόγο σχετικά με την ειδική μου έκθεση, δεν είναι και κάτι που θα ήθελα να το κάνω πολύ συχνά η παράληψη θεσμικών οργάνων να ακολουθούν τις συστάσεις του διαμεσολαβητού θα έπρεπε να είναι σπάνιο γεγονός. Οι εκθέσεις που έχουν κάνει οι προηγούμενοι, οι προκάτοχοί μου δηλαδή, δείχνουν και την προχωρημένη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμών. Ως πολιτικό όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι βεβαίως κυρίαρχο για το τι θα πράξει μετά από την ειδική έκθεση του διαμεσολαβητού. Εγώ επιζητώ την υποστήριξη εκθέσεώ μου, αλλά από εκεί και πέρα είστε ελεύθεροι να πράξετε ό,τι επιθυμείτε. Το θέμα που θα σα θέσω υπόψη σήμερα απαιτεί την ειδική προσοχή του Κοινοβουλίου. Η Frontex, το όργανο, το ευρωπαϊκό όργανο δηλαδή, που έχει ως ρόλο να ενισχύει τι χώρε μέλη για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, δεν δέχθηκε να, την σύστασή μου να ε, δημιουργήσει σύστημα διαχείρισης παραπώνων εσωτερικό. Εγώ δεν λέω ότι αυτό θα έλυνε τα περίπλοκα προβλήματα μετανάστευσης που βρίσκονται στην καρδιά του προβλήματος, αλλά τουλάχιστον θα ήταν ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ε, τήρησης του επίπεδου προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ευρώπη που θεσπίζει ιδίω ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων που η Frontex όπως και κάθε άλλο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ή οργανισμός σε αυτό υπάγονται. Γνωρίζω ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι κάτι το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω δει και το σχετικό βίντεο για τις ε, εκλογές του 2014 που δείχνει και μια εικόνα ενός νεαρού Αφρικανού άντρα που πηδά από ένα σκάφος στα σκοτεινά και παγωμένα νερά. Για να δείξει ακριβώς ποια είναι η ανθρωπιστική πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι ζούμε εν ασφαλεία μέσα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προηγούμενο μήνα 360 άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά πνίγηκαν ε, ε, λίγο έξω από τη Λαμπεντούσα. Πολλοί από εμά συνδέουμε την Λαμπεντούσα με το θαυμάσιο μυθιστόρημα του ε, Ιταλού ε, συγγραφέα γατόπαρδο, που δείχνει την παρακμή μια αριστοκρατική οικογένεια του 19ου αιώνα στην Λαμπεντούσα. Όμω σήμερα η Λαμπεντούσα ίσω δείχνει τον αγώνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που οδηγούν στην απώλεια τόσων ζώων, ακόμη και παιδιών. Τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι έχουν χαθεί τα τελευταία 20 ε, χρόνια σε μια προσπάθεια να φτάσουν τις ε, ευρωπαϊκές ακτές και πόσοι άλλοι άραγε έχουν χαθεί στις θάλασσες που ίσως να τους θυμούνται μόνο οι οικογένειές τους στις πατρίδες τους. Ο πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είπε ότι η Λαμπεντούσα πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής και αυτό είναι ο πυρήνας της σημερινής μου ειδική έκθεσης. Η Frontex δεν δέχτηκε την σύστασή μου, την οποία έκανα μετά από διαρεύνηση των ε, παραπώνων για την τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ιδίω ε, των διατάξεων του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ωστόσο, έλαβα άψογη συνεργασία από την ίδια την Frontex, αυτό το σημειώνω, και το κενό ε, στο θέμα αυτό δεν είναι και τόσο μέγα ώστε να μην μπορεί να καλυφθεί με την ενεργό δράση του Κοινοβουλίου εφόσον αυτό επιλέξει. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παράνομες είσοδοι αποτελούν βεβαίω μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφαλώς και προκαλούνται εντάσει ανάμεσα στο θεμητό συμφέρον ελέγχου της μεταναστεύσεως και από την άλλη μεριά της ανθρωπιστική απέτηση προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Frontex σε συνεργασία με τις χώρες μέλη πρέπει να επιδιώξει να επιτύχει μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στα δύο αυτές αντιφατικές απαιτήσεις. Ο κανονισμός του 2011 επιβάλλει στην Frontex να δρά μέσα στα πλαίσια του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ε, δράση της και να προβλέπει διοικητικές δραστηριότητες για να παρακολουθεί και καταγγελίες που γίνονται στη βάση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και εδώ υπάρχει και ο κώδικας συμπεριφοράς της Frontex που θεσπίζει και ειδικό αξιωματούχο της Frontex για να λαμβάνει παρόμοια παράπονα. Όλα αυτά είναι καλοδεχόμενα βήματα προς τα εμπρός. Τον Μάρτιο του 2013 ο καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος, τότε Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, άρχισε μια πρώτη έρευνα για την πρόοδο που είχε επιτελέσει η Frontex προς την κατεύθυνση ε, ασκήσεως των καθηκόντων αυτών. Διαπιστώσαμε ότι η Frontex επιτελεί πρόοδο για την ε, άσκηση των δραστηριοτήτων που τις επιβάλλει ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ωστόσο, η Frontex δεν διαθέτει μηχανισμό για να αντιμετωπίζει ορθά και να χειρίζεται καταγγελίες παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έλλειψη τέτοιου μηχανισμού σημαίνει ότι η Frontex δεν μπορεί να γνωρίζει πλήρως τις ανησυχίες και τις καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια λειτουργεί. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παράπονα και επομένω κάνουν καταγγελίες δεν έχουν τη δυνατότητα να ακουστούν αμέσως από την Frontex. Το αποτέλεσμα είναι άμεση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών που εφόσον συμβαίνουν παραμένουν ε, άγνωστες. Η Frontex πρέπει να φτιάξει ένα μηχανισμό που θα αντιμετωπίζει τα, τις καταγγελίες των ανθρώπων αυτών των οποίων παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Frontex ωστόσο αποφάσισε να μην δεχτεί τη σύσταση αυτή. Η Frontex λέει ότι με μονομένα επεισόδια τα οποία αποτελούν το αντικείμενο τέτοιων καταγγελιών εν τέλει είναι ευθύνη της χώρας μέλους στην επικράτεια της οποίας συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο οργανισμός δεν έχει άμεση ευθύνη όπως περιγράφεται και ε, το, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ε, μια δύσκολη δηλαδή, ένα δύσκολο πλαίσιο συνθήκων. Εγώ δεν δέχομαι ωστόσο ότι η Frontex δεν φέρει ευθύνη για την δράση προσωπικού που δρά κάτω από την σημαία της. Μπορεί ορισμένες φορές την ευθύνη να την μοιράζεται με την επιμέρους χώρα μέλος, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν φέρει ευθύνη τα μέλη του προσωπικού της συμμετέχουν σε επιχειρησιακές δραστηριότητες ε, στο πεδίο και δεν μπορώ να δεχτώ ωστόσο ότι ο επιμερισμός ευθυνών δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρος. Είναι γεγονός ότι διατίθενται αξιωματούχοι στις ε, περιπτώσεις συνόρων όπου συνεργάζονται με αξιωματούχους της Frontex. Όσοι υφίστανται τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων της Frontex θεωρούν ότι όποιος φέρει το επιβραχιόνιο της Frontex είναι μέλος της Frontex. Οι άνθρωποι αυτοί συνήθως τελούν σε κατάσταση στρες και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Τα είδαμε και τις τελευταίες εβδομάδες τα περιστατικά αυτά και δεν είναι δυνατόν να αναμένει κανείς από ένα απεγνωσμένο άτομο ο οποίο βρίσκεται σε ε, τραγική κατάσταση να μπορέσει να αντιληφθεί την περίπλοκη αυτή ε, διαδικασία καταμερισμού ευθυνών. Είναι λογικό οι άνθρωποι να θεωρήσουν ότι η Frontex είναι ο πρώτο, το πρώτο βήμα στο οποίο μπορούν να καταγγείλουν παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Κάθε άνθρωπος ο οποίος λοιπόν λειτουργεί υπό επίσημη ιδιότητα και φέρει περιβραχιόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει τουλάχιστον μαζί με την χώρα μέλος να είναι υπεύθυνο απέναντι, υπόλογος απέναντι στα ευρωπαϊκά όργανα και μεταξύ αυτών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εν όψη του ιστορικού της καταστροφής της Λαμπεντούσα, της τραγωδίας της Λαμπεντούσα και άλλων α, τέτοιων καταστροφών είναι σημαντικό η Frontex να μπορεί να διαχειρίζεται, αν δέχεται και να διαχειρίζεται άμεσα τα, καταγγελίε των μεταναστών ή άλλων που ζητούν άσυλο. Τον Απρίλιο του 2013 το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε ψήφισμα που ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει ότι οι χώρες μέλη της και η Frontex συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και επομένως θεσπίζουν και σύστημα διαχείρισης καταγγελιών. Τι μορφή μπορεί να έχει αυτό. Για ένα παράδειγμα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που δέχτηκε με την ενθάρρυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να φτιάξει ένα μηχανισμό για πρόσωπα τα οποία επηρεάζονται από έργα που χρηματοδοτεί η ίδια. Λειτουργεί καλά ο μηχανισμός αυτός και έχει βελτιώσει πολύ τη φήμη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα είναι προς το συμφέρον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η Frontex να συμφωνήσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό πρώτης γραμμής. Γνωρίζω ότι ο επικεφαλής του μηχανισμού της ΕΤΕ, κ. Φέλες Μίνο, είναι παρόν και στη διάθεσή σας για να απαντήσετε σε ενδεχόμενες ερωτήσεις που ίσως θελήσετε να του υποβάλλετε για το μηχανισμό αυτό. Ολοκληρώνοντας σήμερα στην πρώτη μου ειδική έκθεση, ζητώ την υποστήριξή σας για να χρησιμοποιήσετε τις εξουσίες που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να απαιτήσετε από την Frontex να θεσπίσει μηχανισμό χειρισμού παραπώνων ώστε όσοι υφίστανται παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους από πράξη ή παράληψη του οργανισμού Frontex να έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν ε, καταγγελίες, να απευθύνουν παράπονα και να γνωρίζουν ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Ράιλι. Ξέρετε ότι το πρωί επικυρώσαμε την απόφαση που πήραν οι συντονιστές μας να προσαρμόσουμε την κατεπίγουσα διαδικασία, να εφαρμόσουμε την κατεπίγουσα διαδικασία για δέκα θέματα πάρα πολύ ευαίσθητα. που αφορούν και τις μεταναστευτικές ροές στην Μεσόγειο και το πρόβλημα της Λαμπεντούζα και τις μεθόδους του Frontex. Θα συνεργαστούμε λοιπόν και θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά στις 16 Δεκεμβρίου. Ξεκινάει η συζήτηση, θα ζητήσω από τους συναδέλφους να είναι πολύ σύντομοι. Ο κύριος Χίγγινς, πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πράγματι σύντομος. Θέλω να καλωσορίσω φυσικά τους συναδέλφους από την Ιρλανδική Βουλή. Πρόκειται για μια εξαιρετική συνάντηση και είμαι πάρα πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο και πράγματι δεν υπήρχε η δυνατότητα να υπάρξει αποζημίωση προς τους ε, αναφέροντες. Ε, έχουμε μια θετική εμπειρία λοιπόν για την κυρία Ράιλι σε εθνικό επίπεδο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που διορίστηκε, επελέγει μάλλον, ως ε, ε, μεσολαβήτρια σε κοινοτικό επίπεδο. Τώρα για τους όρους αναφοράς της Ιρλανδικής Επιτροπή και το άρθρο 11 λέγει ότι ε, μπορεί να συνδιαλέγεται με την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε σχέση με το θέμα της πρωτοβουλίας του Ευρωπαίου Πολίτη, της συλλογής υπογραφών δηλαδή. Έχει σημασία λοιπόν να συνδέσουμε το τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο με το τι συμβαίνει σε ε, ε, επίπεδο κοινοτικό. Η κυρία Ραϊλή έχει δίκιο όταν λέει ότι είναι ένα πολύ σπάνιο συμβάν μια ειδική έκθεση. Δεν πρέπει να είναι πάνω από μία κατέτος και επέλεξε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα με την έκθεση που μας παρουσίασε σήμερα. Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα είναι η ζωή και ο θάνατος. Ξέρετε ότι υπάρχουν χιλιάδες οι οποίοι χάνονται σε αιτήσια βάση και δεν αναφέρεται η απώλειά τους, η θάνατή τους, δεν είναι μόνο στη Λαμπεντούζα. Να πω λοιπόν ότι πράγματι είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός των ε, θεμητών προσπαθειών ελέγχου της μετανάστευσης και της προστασίας των πολιτών και συνεχίζει η κυρία Ρέιλι λέει ότι δεν υπάρχει μηχανισμός στο Frontex σχετικά με τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. και ότι πάρα πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις δεν εντοπίζονται και δεν αναφέρονται και φυσικά δεν επιλύονται. Εμείς σας υποστηρίζουμε κυρία Ρέιλι να υποστηρίξετε κι εσείς με τη σειρά σας ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγξει το Frontex και να δημιουργήσει έναν μηχανισμό παραπώνων από πλευράς του οργανισμού αυτού. Ελπίζω κάτι τέτοιο να συμβεί. Ευχαριστώ. Έχουμε 7 λεπτά στη διάθεσή μας μόνο και έχουν ζητήσει 7 συνάδελφοι το λόγο. Και πρέπει φυσικά να δώσουμε και την δυνατότητα στην κυρία Ράιλι ε, να απαντήσει. Γι' αυτό παρακαλώ ένα λεπτό ο καθένας. Κυρία Γκόντς. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνο και θα είμαι και εγώ πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την ειδική έκθεση που μας παρουσιάσετε. Είμαι ε, μία από τις αντιπροέδρους της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ και πραγματικά ε, στην Επιτροπή μας έχουμε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα ήδη από την αρχή των μεταναστευτικών ροών στην Μεσόγειο γιατί θεωρούμε ότι είναι πραγματικά ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει στην ε, Μεσόγειο. Δεν αναφερόμαστε μονάχα ε, στο κατά πόσον γίνονται ε, σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προφανώς όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό καταγράφεται πολύ αρνητικά στη συνείδηση όλων των Ευρωπαίων. Είναι απολύτως απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα σύστημα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι μεμονωμένες αναφορές, τα μεμονωμένα παράπονα ή καταγγελίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Όκεν. Σας καλωσορίζω θερμά. Κρίμα, κρίμα που δεν ε, μπορέσαμε να σας καλωσορίσουμε επισήμως στην Ολομέλεια. Θα έπρεπε να το είχαμε πράξει. θα μπορούσε ενδεχομένως η κυρία Μασόνη να ε, το ζητήσει βεβαίως ε, ως πρόεδρος της Επιτροπής. Εν περιπτώσει Έχω πολλά ζητήματα να συζητήσω ε, μαζί σας, αλλά δυστυχώς όπως είπε και η Πρόεδρος δεν έχουμε χρόνο. Το μόνο που θα πω είναι ότι ενδεχομένως τα πλαίσια της Frontex ε, και θα πρέπει να μπουν και οι ετούντες ε, άσυλο, αλλά κυρίως μια πολύ σημαντική ομάδα αυτή των Παλαιστινίων που τους φέρονται σαν να είναι σκουπίδια. Ε, και συνήθως δεν τους παρέχεται άσυλο ε, και τους ξαναστέλνουν ε, στο στόμα του λύκου. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που είναι απάτριδες στην ουσία δεν έχουν που να πάνε. Αναφέρομαι και σε μια υποκατηγορία που είναι πολύ σημαντική, τα παιδιά ε, τα οποία βρίσκονται στις, στα σύνορα των χωρών μας ε, χωρίς γονείς. Ε, ασυνόδευτα λοιπόν παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση. Πρέπει να πω ότι όλοι υφίστανται κακομεταχείριση αλλά οι Παλαιστίνοι ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ κύριο Γάλλο. Ευχαριστώ και εγώ πραγματικά όσο γίνεται συντομότερα. Κυρία Ρέιλι, σας ευχαριστώ που προσήλθατε για την, για την ειδική έκθεσή σας. Είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα, όντως διότι υπάρχει και σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Η πρώτη καλή είδηση είναι ότι η Επιτροπή Αναφορών στο σύνολό της διακομματικά δέχθηκε την έκθεσή σας και επιθυμεί να τη συζητήσει. Και όχι μόνο. Θεωρούμε ότι οφείλουμε να ε, συζητήσουμε την έκθεσή σας. Η Ευρώπη ως οργανισμός δικαίου και δημοκρατίας, σε αυτά εντάσσονται βεβαίως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα κάποιος να μπορεί κάπου να αναφέρεται, να υποβάλει ένα παράπονο. Όπως είπα η Επιτροπή Αναφορών θα εγγύψει στο θέμα εντατικά. Η δική μου ερώτηση προς εσάς, ή μάλλον θα ήθελα πρώτα να πω, ότι δεν μπορούμε να καταστήσουμε τη Frontex υπεύθυνη για τα πάντα πρέπει. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε και όταν σημειώσουμε κάποιο έλλειμμα να φροντίσουμε να καλυφθεί. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα σημαίνει βεβαίως αυτό ότι σε αυτά περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να υποβάλει κανείς καταγγελία. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πού είναι το πλέον απλό και αποτελεσματικό να εγκαταστεί ο μηχανισμός υποδοχής των ε, καταγγελιών. Ε, Um, Μέρφυ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω την κυρία Ρέιλ. Είναι πάρα πολύ θετικό που έχουμε αυτήν την πρώτη ε, παρουσίαση της ειδική ε, ε, έκθεσης. Πρέπει όμως να κάνω ένα παράπονο την προηγούμενη εβδομάδα ε, είχαμε την ε, ανάπτυξη ενός μεγάλου χαρτιού με χιλιάδες υπογραφές ε, ανθρώπων οι οποίοι χτύπησαν στις πόρτες αυτού του οχυρού της Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι ένας λόγος για να σταματήσουμε πια αυτήν την φρουριοποίηση της Ευρώπης, αυτήν την στρατιωτικοποίηση ε, της ε, ε, Ευρώπης και η Frontex συμμετέχει βέβαια στη διαδικασία αυτή, θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Η Frontex βέβαια προσπαθεί να λειτουργήσει στα πλαίσια ενός νομικού κοινού ανάμεσα τις αρμοδιότητες τι ενωσιακές από τη μία πλευρά ε, και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών που επισήμω είναι αρμόδια ε, για το ε, ζήτημα. Πάντω στηρίζω την πρόταση ε, να υπάρξει ένας ε, κανονικός μηχανισμός ελέγχου στα πλαίσια της ε, Frontex. Εγώ βεβαίως προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να διαγραφεί η Frontex, να διαλυθεί το φρούριο της Ευρώπης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε πια αυτήν, την, αυτά τα λόγια, τα περιτά μόνο για, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να περάσουμε στις πράξεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζανώστικα. Πολύ σύντομα. Κυρία Ρέιλι. Λέτε ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ζητά την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και εμείς ζητούμε ε, την ε, δική σας ε, στήριξη. Ζητούμε λοιπόν ε, να μας πείτε εάν ε, θα πάτε και στην Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ, είμαι μέρος και αυτής της Επιτροπής και πραγματικά θα ήθελα να σας ζητήσω, αν δεν το έχετε πράξει μέχρι τώρα, να παρουσιάσετε την έκθεση αυτή για τη Frontex και στη ΛΥΜΠΕ, η οποία είναι η καθήλυνα αρμόδια για τη Frontex. Uh, Καλά. Ολοκληρώθηκε εδώ η συζήτηση. Μπορώ να επανέλθω λοιπόν στην κυρία Ορέιλη ώστε να μπορέσει να απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλες και όλους για τις παρεμβάσεις σας. Τσέν και σε σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Κύριε Άουκεν, α, βλέπω ότι ήταν υποχρεωμένο να αποχωρήσει. Βεβαίως ε, δέχομαι το σχόλιο για τους Παλαιστινίους. Ομάδες όπως και Παλαιστίνοι που προέρχονται από τη Συρία προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ολόκληρη η αξία του μηχανισμού υποβολής παραπώνων είναι ότι θα επιτρέψει στο ίδιο το όργανο πώς, να δει πώς λειτουργούν οι διαδικασίες του. Έχοντας συζητήσει και με τον κύριο Αλκάρπε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει να σας πει και εσάς αυτά που είπε και σε μένα, ότι η εισαγωγή του μηχανισμού υποβολής παραπώνων θα ωφελήσει και, το ίδιο, και τον ίδιο τον οργανισμό, εν προκειμένου την Frontex. Νομίζω ότι η Frontex θέλει να βελτιωθεί ως οργανισμός. Θέλει να αρθεί στο ύψος του ε, ορθού επίπεδου προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όπως είπα και στις αρχικές μου παρατηρήσεις, η Frontex δεν θεωρεί ότι φέρει την ευθύνη αυτή για τα όσα είπε ο κύριος Γιάρο ότι δεν μπορεί κανείς να φορτώσει όλες τις ευθύνες στην Frontex, αυτό είναι απόλυτα σωστό. Ωστόσο η αξία του μηχανισμού είναι ότι μέσα από την ανάλυση του παραπόνου θα μπορέσουν να κατανοήσουν και οι υπεύθυνοι πού στην ευχή βρίσκεται η συγκεκριμένη ευθύνη. Αυτό νομίζω ότι είναι η αξία της ιδέας. Ο Πολ είπε μερικά σχόλια πρόκειται βεβαίω για τεράστια πολιτικά θέματα τα οποία εμπλέκονται εδώ. Και πάλι νομίζω ότι η αξία του μηχανισμού υποβολής παραπώνων είναι ότι ανοίγει τις εσωτερικές διαδικασίες ενός οργανισμού ώστε και από μέσα και απ' έξω να μπορούν να δουν πώ λειτουργεί, πώς υποτίθεται ότι πρέπει να λειτουργεί και βεβαίω και σε σχέση με με τα πρότυπα ε, σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όσον αφορά την ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει ακριβώς. Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως δέχομαι προσκλήσεις από οποιαδήποτε κοινοβουλευτική επιτροπή ε, να εμφανιστώ ενώπιον της. Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως η Επιτροπή Αναφορών θα ζητήσει γνωμοδοτήσεις από άλλες επιτροπές. Οτιδήποτε μπορώ να πράξω για να συμβάλλω στις, στον προβληματισμό σας εγώ πολύ ευχαρίστω θα το πράξω. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ωρέλη και ευχαριστώ επίσης και όλους και όλες και όλους τους ευρωβουλευτές στο πνεύμα συνεργασίας που δείξατε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε έγκαιρα. Ευχαριστώ και τις και τους διερμηνείς που μας δώσαν πέντε λεπτά παραπάνω και εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας συνεδρίαση.